Uh, Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Οι πράσινοι ζήτησαν να προσταθεί μια προφορική ερώτηση για διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς την κατάσταση των πραγμάτων των εξή ε, θεμάτων. Πρόσβαση σε περιβαλλοντικά θέματα, την βιώσιμη ανάπτυξη, την επιστηστική ασφάλεια την επισήμανση και τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Αυτό το προβλέπουμε ως νέο σημείο 17α την Τετάρτη το απόγευμα. Μετά, αργότερα, έχουμε Αμέσως μετά το σημείο είναι οι ανακοινώσεις του Προέδρου. Η πρώτη ανακοίνωση είναι οι επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής. Επειδή συμπίπτουν με τις ακροάσεις των υποψήφιων επιτρόπων, η συνεδρίαση η και 30 η Σεπτεμβρίου καθώς και 6 και 7 η Σεπτεμβρίου αναβάλλονται. Οι ακροάσεις της Επιτροπής ΕΜΒΗ θα λάβουν χώρα ως εξής. Ακρόαση του Επιτρόπου Βέλα μαζί με την Επιτροπή Αλίας. Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στις 2.30. Ακρόαση του κυρίου Αντρίου Κάιπης, 3η 30 Σεπτεμβρίου στις 9. Ακρόαση του κυρίου Κανιέτε μαζί με την Επιτροπή Ήτρε, Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, στις 6. Ακρόαση της Αντιπροέδρου Μπράτουσεκ μαζί με την Επιτροπή Ήτρε την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 2.30. Τα μέλη θα λάβουν προσκλήσεις και τα σχέδια μερίσες διάταξης από την ε, ε, Γραμματεία μαζί με το πρόγραμμα των ακροάσεων. Ιδίω για αυτέ ε, τι επιτροπέ τη ακροάσεων όπου συμμετέχει η επιτροπή μα. Δεύτερον ανακοίνωση, δεύτερη ανακοίνωση από μένα. Συνάντηση στις 10, στις 30 μάλλον Σεπτεμβρίου, για να συζητήσουμε το, την αναδιατύπωση του ΣΕΤΙΣ του ΣΥΤΙΣ μάλλον. Θα το συζητήσουμε με την Ιταλική Προεδρία, γιατί υπάρχει εδώ ε, μπλοκάρισμα του θέματος λόγω διαφωνίας ε, Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για τις κατεξοδότηση πράξεις. Θα προσπαθήσουμε να εξεύρουμε μία λύση. Έπειτα ανακοίνωση για την διερμηνία, η οποία διατίθεται σε 21 γλώσσες σήμερα. Λυπούμεθα για τα εστονικά και για τους συναδέλφους από τη Μάλτα, αλλά δεν θα έχουμε διερμηνία για αυτούς. Από τη γλώσσα τους. Ως συνήθως, τα πρακτικά διατίθενται από την εφαρμογή e-meeting και επίσης θα μεταδοθεί στο διαδίκτυο συνεδρίασή μας. Άλλη ανακοίνωση για την ψηφιακή υπογραφή οι συνάδελφοι έχουν στη διάθεσή τους την εφαρμογή ηλεκτρονική υπογραφή που επιτρέπει την υποβολή ε, τροπολογιών με PIN ή smart card η ηλεκτρονική υπογραφή θα έχει πολλά ωφέλη ως προς την κινητικότητα, την ασφάλεια και την έγκαιρη υποβολή των τροπολογιών καθώς και τη διαχείρισή τους. Προκειμένου να αξιοποιήσετε την εφαρμογή αυτή, Digital Signature, θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση επισήμως για PIN ή για Smart Card ή για έξυπνη κάρτα. Η πρώτη χρήση της ε, ε, επιλογής αυτής, της εφαρμογής αυτής, θα ξεκινήσει δοκιμαστικά στη συνεδρίαση της 9 η Οκτωβρίου στις 4, στις 6. Ε, τώρα, για την εφαρμογή e-meeting, για να μειώσουμε την κατανάλωση χάρτου, το άνευ χάρτου πρόγραμμα του Κοινοβουλίου με την εφαρμογή e-meeting δίνει τη δυνατότητα να δείτε όλες, όλα τα έγγραφα μιας συνεδρίας της Επιτροπής μέσω ταμπλέτας ή λάπτοπ. Γι' αυτό προσκαλέσαμε δύο συναδέλφους της Γενικής Διεύθυνσης ITEC να μας παρουσιάσουν την εφαρμογή αυτή και τους προσκαλώ να μας κάνουν μια σύντομη παρουσίαση για να μας εξηγήσουν πώς θα λειτουργήσει. Thank Έχετε το λόγο. Uh, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να σας παρουσιάσουμε την εφαρμογή e-meeting, electronic meeting Ορισμένοι εξημών, από την προηγούμενη θητεία δηλαδή, τα έχετε ακούσει τα σχετικά και ίσως μάλιστα να έχετε χρησιμοποιήσει και το e-meeting, επειδή όμως σίγουρα υπάρχουν πολλοί νέοι ευρωβουλευτές αλλά και μέλη του προσωπικού, θα είναι καλό να σας εξηγήσουμε πώς λειτουργεί. Όπως είπε ο πρόεδρος σας, το e-meeting έχει σκοπό να συμβάλλει στη μείωση του χαρτιού που καταναλώνει το Κοινοβούλιο. Πολύ χαρτί τυπωνόταν, ιδίω για τις συνεδριάσεις. Λίγοι όμως χρησιμοποιούσαν όλο αυτό το χαρτί. Όλα αυτά τα έγγραφα, δηλαδή τα τυπωμένα έγγραφα. Αυτό οδηγούσε σε πολύ σπατάλη. Το e-meeting πάει να αντικαταστήσει το χαρτί βέβαια, αλλά ταυτόχρονα και να συμβάλλει στην αποδοτικότερη εργασία όλων. Όχι μόνο στις αίθουσες συνεδριάσεων και στα γραφεία, αλλά και αλλού, μέσω των κινητών συσκευών. Πρόκειται λοιπόν για εφαρμογή δική μας, την οποία εξελίξαμε εμείς, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο εργασία του Ευρωκοινοβουλίου. Είναι διαθέσιμο σε όλα τα tablet, λάπτοπ, FE τηλέφωνα, είτε έχετε 3G, είτε 4G κλπ. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σαν να είναι χαρτί. θα κάνουμε μια παρουσίαση του e-meeting και όσοι έχετε τέτοιες συσκευές μαζί σας, τάμπλετ ή εφή τηλέφωνα, μπορείτε να τα δείτε. Έχουμε διανύμει μία σελίδα, έναν οδηγό μια σελίδος για να σας εξηγήσουμε πώς λειτουργεί αυτό το e-meeting. Δεν θέλουμε βέβαια να διανύμουμε και πολύ χαρτί για το project αυτό, αλλά είναι μια εξαίρεση. Σύντομα λοιπόν, πρόκειται για εφαρμογή web, άρα χρειάζεται να έχετε, μια, να έχετε την διεύθυνση, την διεύθυνση web που τη βρίσκεται πάνω στην σελίδα που σας δώσαμε και χρειάζεστε βέβαια και τα διαπιστευτήριά σας, login και password. Με την άδειά σας να παρακαλέσω τον συνάδελφό μου να κάνει μια σύντομη παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας του e-meeting και βέβαια αν θέλετε μετά θα σας απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ, καλημέρα. Θα σας τα δείξω σε iPad, που μπορείτε όμως να χρησιμοποιήσετε και άλλα σχετικά μηχανήματα. Το e-meeting λοιπόν είναι εφαρμογή του δικτύου. Δεν χρειάζεται δηλαδή να εγκαταστήσετε λογισμικό. Για να έχετε πρόσβαση θα πάτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωκοινοβουλίου και μετά θα βάλετε κάθετος ή meeting. Είναι εσωτερική βέβαια η εφαρμογή αυτή. Επομένως πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα διαπιστευτήριά σας, δηλαδή username κλπ. Και αυτό είναι και το ε, συνθηματικό μου, το password. Once the Όταν θα έχετε για πρώτη φορά πρόσβαση στην εφαρμογή, θα έχετε αυτό το πρώτο, την πρώτη σελίδα. Διαλέγετε λοιπόν τη γλώσσα, την επιτροπή και την ημερομηνία. Πατάω το start και αυτό είναι το interface που βλέπετε. Στις διάφορες γλώσσες βέβαια, έτσι, όχι μόνο στα γαλλικά. Και διαθέσιμες στην ίδια interface είναι και όλες οι κοινοβουλευτικές επιτροπές. Μπορώ να κάνω και ένα zoom in, μια μεγέθυνση δηλαδή, για να δείτε πού χτυπάω. Βλέπετε λοιπόν εδώ τα αγγλικά. Και μετά πάει εκεί, πάτε εκεί που λέει choose, επιλογή δηλαδή, της Επιτροπής και ψάχνω και βρίσκω την environment, περιβάλλον δηλαδή. Συνολική τώρα ε, άποψη, αριστερά είναι το, η συνάντηση και δεξιά είναι η μερίσια διάταξη της κάθε μιας συνάντησής σας. Επάνω δεξιά τώρα βλέπετε τις διάφορες παραμέτρους για την πρόσβαση. Βλέπετε για παράδειγμα την ημερήσια διάταξη. Μπορώ να πάω μετά στα documents, έγγραφα. Θα σας πω μετά και εκεί που λέει η committee. Έχω το λεγόμενο feedback, αν θέλετε κάτι καινούριο ή αν θέλετε βοήθεια. Και τέλος έχετε και τη βοήθεια, η οποία σας εξηγεί αυτόματα πώς λειτουργεί η εφαρμογή. Εδώ έχουμε το appendix, μπορείτε όμως να βρείτε και κάθε έγγραφο εκεί και τα τελευταία πιο πρόσφατα δηλαδή που έχουν αναρτηθεί στο εσωτερικό διαδίκτυο. Επίσης εδώ έχετε και τρόπο να βρείτε ένα θέμα της ημερήσιας διάταξης που μπορείτε να το στείλετε μετά σε ένα συναδελφό σας ή στο συνεργάτη σας. Με περισσότερες λεπτομέρειες τώρα το περιεχόμενο της εφαρμογής. Αν θέλετε δηλαδή από αριστερά να διαλέξετε τη σημερινή συνεδρίαση, 24η δηλαδή, 9 δεξιά θα δείτε ενημερωμένη την ημερήσια διάταξη με όλα τα σχετικά έγγραφα. Εκεί που έχει ένα συν βλέπουμε έξτρα πληροφορίες για κάθε συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με έξτρα information δηλαδή βέβαια για τον εισηγητή και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τυπώνονταν πριν. Η ιδέα λοιπόν είναι να μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή e-meeting για να υποκαταστήσει όλο αυτό το χαρτί που τυπώνεται ακόμη τώρα. Για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως βλέπετε και το συνδεδεμένο έγγραφο. Εδώ για παράδειγμα μπορώ να δω το σχέδιο ημερησίας διατάξεως σε όποια γλώσσα θέλω. Ρουμανικά για παράδειγμα εδώ βλέπετε ξαφνικά να εμφανίζεται το έγγραφο στα ρουμανικά. Αν θέλω τώρα να δω, να κάνω μια προσθήκη, μπορώ να το ανοίξω σε άλλη εφαρμογή. Θα εξαρτηθεί από το τι είδους editor έχετε ε, στο μηχάνημά σας. Εδώ το ανοίγω στο Adobe Reader. Αυτός ο editor λοιπόν είναι διαθέσιμος στο μηχάνημα που έχω μπροστά μου. Εδώ μπορώ να κάνω interact με το έγγραφο, βλέπετε κάνω ένα κύκλο, μπορώ να κάνω μια σημείωση. Να βάλω ένα σχόλιο. οτιδήποτε κάνω είναι local, είναι μόνο τοπικό, δηλαδή δεν πηγαίνει σε κανέναν άλλο. Οποιαδήποτε σημείωση και οτιδήποτε άλλο κάνω στο έγγραφο αυτό. εφόσον τελειώσω τις σημειώσει μου κτλ. μπορώ να μοιραστώ το έγγραφο αυτό, να το στείλω δηλαδή σε συνεργάτη μου ή στο, σε άλλο βουλευτή κτλ. Και ό,τι έχω κάνει αποθηκεύεται και στη νέα αυτή εκδοχή του κειμένου μου, την οποία μπορώ να στείλω κι αλλού. Ένας λοιπόν τρόπος να χρησιμοποιήσω το e-meeting. Μπορώ να ξαναδώ ανα πάσα στιγμή το έγγραφο όλες τις γλωσσικές εκδοχές, μπορώ να ανοίξω το έγγραφο, μπορώ να κάνω interact μαζί με το έγγραφο δηλαδή, να, ε, να δράσω επ' αυτού και μπορώ να το μοιραστώ και με άλλους. Τώρα έχουμε και μια άλλη εφαρμογή και με την ευκαιρία αυτή να σας πω, που είναι η e-committee, e-committee, όχι πλέον e-meeting, εδώ αυτό είναι το εργαλείο για κάθε επιτροπή. Ένας χώρος όπου κάθε επιτροπή μπορεί να αποθηκεύσει έγγραφα που έχουν σχέση με τις εργασίες της. Μπορείτε να βρείτε δηλαδή έξτρα πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν στην προπαρασκευή σας για την ε, συνάντηση. Έχετε σχέδια εκθέσεων, σχέδια γνωμοδοτήσεων, τροπολογίες, καθώς και τις σχετικές προθεσμίες για την υποβολή τους. Αυτή είναι η e-committee. E πολύ σύντομα εδώ σε μια οθόνη. Ο χώρος αυτός είναι πιο εκτεταμένος, είναι πλουσιότερος. Εδώ έχετε την mobile view σε οποιοδήποτε δηλαδή κινητή συσκευή και με οποιαδήποτε ε, διευκρίνηση οθόνης. Έχω λοιπόν εδώ όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα μέλη τους συνεργάτες, πληροφορίες πώς θα έλθω σε επαφή με τους συνεργάτες, με πολιτικές ομάδες, με τους ε, βοηθούς και ούτω καθεξής. Αυτή λοιπόν είναι η e committee, ε committee. Και το e-meeting σας το έδειξα πριν. Εδώ ολοκληρώνεται η παρουσίασή μου και αν έχετε ερωτήσεις, πολύ ευχαρίστως να σας απαντήσω. Ο πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Δεν νομίζω να υπάρχουν ερωτήσεις ή απορίες. Και απλώς με την παρουσίαση αυτή θέλαμε να δείξουμε στους συναδέλφους ποια είναι τα εργαλεία που έχουμε στη θέση μας. Και θα φροντίσουμε με την ε, Γραμματεία και την Γενική Διεύθυνση ITEC να οργανώσουμε συγκεκριμένη συνάντηση για τους βοηθούς, για να εκπαιδευτούν και να προωθηθεί χρήση όλων αυτών των ηλεκτρονικών εργαλείων. Ευχαριστώ τη Γενική Διεύθυνση ITEC και θα έλεγα να περάσουμε αμέσως στην ε, σειρά της ημερήσιας διάταξης. Επόμενο σημείο, το σημείο 4 μετά την τοποθέτηση του Συμβουλίου για τη δυνατότητα των κρατών μελών να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στην επικράτειά τους. Κατόπιν λοιπόν της ε, τοποθέτησης του Συμβουλίου επί του θέματος θα περιοριστώ να θυμίσω πόσο το θέμα αυτό έχει μια μακρά πορεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την αρχική της πρόταση το 2010, το Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2011 κιόλας τοποθετήθηκε σε πρώτη ανάγνωση και μόλις τον Ιούνιο του 2014 επετέχθη πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο με ευνοϊκή ψήφο από όλα τα κράτη-μέλη με εξέρεσε το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο που απήχαν. Στα τέλη Ιουλίου στις 23 το Συμβούλιο ενέκρινε την επίσημη τοποθετησή του η οποία απεστάλλει για έγκριση στην Ολομέλεια στις 15 Σεπτεμβρίου. Επειδή η Ιταλική Προεδρία θέλει να αποπειραθεί την επίτευξη συμφωνίας σε δεύτερη ανάγνωση πριν το τέλος του 2014 έχουμε καθορίσει το εξής χρονοδιάγραμμα. 13 Οκτωβρίου. Σχέδιο έκθεσης. Θα το συζητήσουμε στην Επιτροπή μας, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 15 Οκτωβρίου. Ψηφοφορία στην Επιτροπή μας για την εντολή 5 Νοεμβρίου και ευχόμενη να επιτευχθεί συμφωνία με το Συμβούλιο έγκριση της συμφωνίας Γενάρη του 2015 και ψηφοφορία στην Ολομέλεια και πάλι τον Ιανουάριο του 2015. Για το σημείο αυτό μόνο αυτές τις πληροφορίες θέλω να σας δώσω για το χρονοδιάγραμμα. Επόμενο σημείο, σημείο 5 έγκριση των πρακτικών της, ε, των προηγούμενων συνεδριάσεων 23 και 24 Ιουλίου και 3 Σεπτεμβρίου του 2014 και οι δύο. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, πριν την λήξη της ε, πρωινής μας αυτής συνεδρίασης, τα πρακτικά θα θεωρηθούν εγκεκριμένα. Και κατόπιν να πάμε στο επόμενο σημείο, ένσταση βάσει του άρθρου 106 για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, ΣΕΔΕ, κατάλογος τομέων και κλάδων οι οποίοι θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα για την περίοδο 2015 έως 2019. Για το σημείο αυτό να πούμε ότι την ένσταση αυτή υπέβαλε η ομάδα των Πρασίνων, του συναδέλφου Eichhout. Του δίνω λοιπόν το λόγο για να μας την παρουσιάσει. Παρακαλώ. Thank you very ε, Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πολύ όλους που είσαστε εδώ για να συζητήσουμε αυτό το θέμα που μας οδήγησε σε ένα σωρό email, ανταλλαγές με lobbyist κλπ. Ας αρχίσουμε. Τι είναι η διαρροή άνθρακα. Έχουμε ένα σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και ξέρουμε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν πρόβλημα με το διεθνή ανταγωνισμό. Οπότε, αν μια επιχείρηση έχει τέτοιο πρόβλημα με το διεθνή ανταγωνισμό, αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι η επιχείρηση αυτή μπορεί χωρίς να πληρώσει, χωρίς το σύστημα πληστηριασμών δηλαδή, να μπορέσει να έχει διαθέσιμες ποσότητες εκπομπών. Να υπάρχει δηλαδή μία εξαίρεση για τις επιχειρήσεις εκείνες που έχουν πρόβλημα με το διεθνή ανταγωνισμό. Εκείνες παίρνουν δωρεάν ε, κατανομή ποσοτήτων. Πώς όμως να υπολογίσουμε ποιες είναι οι επιχειρήσεις που μπορούν να έχουν τέτοια δωρεάν κατανομή, είναι ένα σύστημα το οποίο ήδη είχε αποφασιστεί από το 2008. Ποιες επιχειρήσεις η μεθοδολογία είναι πάρα πολύ βέβαια περίπλοκη, γίνονται υπολογισμοί και καταλήγουμε στο θέμα αυτό της διαρροής άνθρακα. Τώρα, το 2009 ήδη εκφράστηκαν διάφορες αντιρρήσεις στην Επιτροπή Περιβάλλοντος όσον αφορά τη μεθοδολογία αυτή, γιατί είπαμε ότι έτσι θα διηγηθούμε σε περιβολικά πολλές επιχειρήσεις που θα εντάσσονται στον κατάλογο για τη διαρροή άνθρακα. Γιατί τελικά όλες περίπου επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κινδυνεύουν να μπουν σε αυτό το κατάλογο. Και αποδεχτήκαμε σωστή, γιατί σήμερα πάνω από 95% των ε, εκπομπών της βιομηχανίας ε, διοξιδίου του άνθρακος βρίσκονται στον κατάλογο αυτό. Δηλαδή πραγματικά αν δεν έχετε μπει σε αυτό το κατάλογο ως βιομηχανία κάτι περίεργο κάνετε. Γιατί τελικά έχουν ενταχθεί λίγο πολύ όλες. Ήδη διαμαρτυρηθήκαμε για αυτό το 2009 αλλά τότε μας υποσχέθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το 2014 θα αναθεωρηθεί ο κατάλογος αυτός. Θα ενημερωθεί και το λέει και η νομοθεσία του 2008 ότι θα πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση. Και από το 2008 μέχρι το 2020 τώρα είναι η στιγμή που μπορεί να υπάρξει αναθεώρηση του καταλόγου αυτού και να βγουν επιχειρήσεις από αυτόν τον κατάλογο. Το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μόνο να προστίθενται επιχειρήσεις μπορεί. Μας το υποσχέθηκαν λοιπόν, είμαστε στο 2014, μέχρι τώρα, επειδή είμαστε στο 2014, περιμέναμε την αναθεώρηση, ήρθε το καλοκαίρι. Έκανε δηλαδή τη δουλειά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήρθε με μία εκτίμηση αντικτύπου. Αυτή η εκτίμηση όμως δυστυχώς δεν είναι δημόσια. Δεν υπάρχει διαφάνεια η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποσχέθηκε καλύτερες ρυθμιστικές διαδικασίες. Ε, λοιπόν, το βασικό θα ήταν τέτοιες μελέτες αντικτύπου να γίνονται ανοιχτές για το κοινό, ώστε να ξέρουμε τι λένε. Βέβαια, Τίποτα δεν μένει μυστικό όπως ξέρετε τελικά να το ψάξει κανείς και το ψάξαμε και το βρήκαμε και το στείλαμε σε όσους πιστεύουμε ότι ενδιαφέρονται γιατί θεωρούμε ότι είναι σημαντικό όλοι να ξέρουμε την έκθεση αυτή αντικτύπου. Το μεγαλύτερο λοιπόν πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι για τον καθορισμό ποια επιχείρηση θα μπει στον κατάλογο αυτό διαρροής άνθρακα και ποιο όχι χρησιμοποιείται μια τιμή 30 ευρώ ανατόνο διοξιδίου του άνθρακα. Και όλοι ξέρουμε ότι η τρέχουσα τιμή είναι περίπου 5 ευρώ. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί όσο πιο ακριβή θεωρείται την τιμή του διοξιδίου του άνθρακα, τόσο πιο πολλές επιχειρήσεις αποδεικνύεται τελικά ότι έχουν πρόβλημα με τον διεθνή ανταγωνισμό. Αν βάζαμε 100 ευρώ, α πούμε, ε, προφανώ όλε οι επιχειρήσει θα έπρεπε να μπουν. Με την υπόθεση δηλαδή του 30% βάζουμε 95% των επιχειρήσεων στον κατάλογο, ότι κινδυνεύουν δηλαδή από τον διεθνή ανταγωνισμό. Είναι πολύ ενδιαφέρον επίσης να δούμε την έκθεση αντικτύπου, γιατί στη σελίδα 33, που πολύ ωραία διατυπώνεται, περιλαμβάνει το πιο ακραίο σενάριο που λέει ότι στην ακραία περίπτωση το 2020 η τιμή θα είναι 12 ευρώ. Οπότε η έκθεση αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της ίδιας λέει 12 ευρώ που σημαίνει ότι δεν είναι λογικό να χρησιμοποιούμε το 30% και για αυτούς που λένε ναι, μα είμαστε υποχρεωμένοι να βάλουμε το 30% γιατί υπάρχει στην νομοθεσία πάλι στη σελίδα 33 λέει, επιλέξει, ότι η οδηγία δεν αναφέρει ότι πρέπει ρητά να χρησιμοποιείται μία τιμή και ότι πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα αντικτύπου για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα βάσει συγκεκριμένων δεδομένων. Τα έχουμε λοιπόν στην έκθεση αντικτύπου. Και το συμπέρασμα της έκθεσης αντικτύπου, στη σελίδα 4, λέει ότι η επιλογή που σημαίνει ότι μπαίνουν λιγότεροι τομείς στον κατάλογο από ό,τι προηγουμένως, θα μειώσει κατά 4,5% για ολόκληρη την περίοδο 2015 μέχρι 2019. Κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε 5 δισεκατομμύρια επιπλέον έσοδα για τις χώρες μέλη. Κάτι άλλο σημαντικό είναι ότι αναφέρεται πως δεν μιλάμε για μια τιμή άθρακα που θα ανέβει ή θα κατέβει, μιλάμε για το θέμα της κατανομής. Τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι μια κατανομή. Ποιος πληρώνει και ποιος παίρνει. Η σημερινή πρόταση της Επιτροπής είναι να κρατήσουμε τα 30 ευρώ, δηλαδή αντιφάσκει εδώ με την ίδια της την έκθεση αντικτύπου και τα χρήματα αυτά πηγαίνουν σε επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόβλημα με το διεθνή ανταγωνισμό, απλώς και μόνο γιατί βρίσκονται σε αυτό το κατάλογο, ο οποίος έχει καταρτιστεί με ιδιαίτερα ψηλή τιμή άνθρακα. Οπότε τι κάνουμε, τα 5 δισεκατομμύρια είναι των φορολογούμενων. Και εδώ θέλω να πω στους συναδέλφους από το ΕΛΚ, οι οποίοι κάθε φορά στις οικονομικές συζητήσεις λένε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί με τα χρήματα των φορολογούμενων. Τώρα συζητάμε αυτό το θέμα και ξαφνικά τα 5 αυτά δισεκατομμύρια για τα οποία πρέπει να πληρώσει ο φορολογούμενος για τη βιομηχανία, που δεν έχει πρόβλημα με το διεθνή ανταγωνισμό, εξαφνικά δεν τους ενδιαφέρουν και βασίζεται και σε λαθασμένα δεδομένα. Δείτε, εγώ δεν λέω να απαλλαγούμε από ολόκληρο τον κατάλογο. Όχι, εγώ λέω να χρησιμοποιήσουμε μια πιο σωστή τιμή άνθρακα για να καθοριστεί ο κατάλογος διαρροής άνθρακα. Η προστασία δηλαδή της βιομηχανίας να γίνει για τις επιχειρήσεις εκείνες που τη χρειάζονται. Αυτό σημαίνει καλύτερη ρύθμιση στο κάτω-κάτω. Καλύτερη νομοθετική ρύθμιση βελτίωση της ανάλυσης και ανάλογες αποφάσεις. Τα χρήματα να πηγαίνουν εκεί που χρειάζονται και όχι να βάζουμε το φορολογούμενο να πληρώνει για βιομηχανίες που δεν τα χρειάζονται γιατί δεν έχουν πρόβλημα με το διεθνή ανταγωνισμό. Έχω απογοητευτεί κυρίως με τον Πίτερ γιατί το ξέρει το θέμα και δεν καταλαβαίνω γιατί το χειρίζεται έτσι όπως το χειρίζεται. Άρα λοιπόν το θέμα είναι η ανακατανομή των χρημάτων. Και έρχομαι στο τελευταίο. Τώρα και φυσικά υπάρχει το λόμπι της βιομηχανίας που λέει «Μα όλα αυτά δημιουργούν αβεβαιότητα στη βιομηχανία». Μα όπως είπα πριν, το 2008 ήδη είχε προβλεφθεί αναθεώρηση για το 2014 και η εκτίμηση δικτύπου δείχνει ότι τα 30 ευρώ δεν είναι κάτι ρεαλιστικό και σωστό. Όλοι λένε ότι πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική τιμή. Και τα κράτη-μέλη. 16 και μισό ανέφερε κάποια στιγμή η έκθεση και έλεγε ότι έτσι θα υπάρξει μια πιο σωστή και δίκαια κατανομή. Η πολιτική απόφαση όμως είναι διαφορετική. Εμείς ως κοινοβούλιο μπορούμε να εκφράσουμε αντίρρηση. Και μάλιστα εγώ θα έλεγα ότι έχουμε την υποχρέωση να εκφράσουμε αντίρρηση ένσταση. Επειδή συναποφασίζουμε, πρέπει λοιπόν να κάνουμε ένσταση και να πούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάνετε σωστή πολιτική. Αυτή εδώ δεν είναι καλύτερη νομοθετική ρύθμιση, αλλά χειρότερη πρέπει να δράσετε βάσει των αποτελεσμάτων και των συμπεράσματων τη έκθεσης αντικτύπου σα. Έχουμε χρέο, δηλαδή, το οφείλουμε ω ευρωβουλευτές να αντιταθούμε, να υποβάλουμε ένσταση και να ζητήσουμε νέα πρόταση. Η βιομηχανία το ήξερε ότι θα υπάρξει αναθεώρηση. Η βιομηχανία το ξέρει ότι έχουμε το δικαίωμα στην ένσταση. Οπότε το μόνο που κάνουμε είναι ότι δρούμε βάσει των δικαιωμάτων που έχουμε Οφείλουμε να το κάνουμε αυτό και να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθουμε σε έναν άλλο κατάλογο διαρροής άνθρακα που τον έχουν και έτοιμο. Αν λοιπόν βάλουν τη σωστή τιμή θα έρθουν με ένα νέο κατάλογο διαρροής άνθρακα και βάσει αυτού να πορευτούμε. Εγώ δεν λέω ότι πολύ μου αρέσει όλη αυτή η δουλειά, αλλά λέω ότι για μένα είναι θεμελιώδες γιατί έχει να κάνει με την ποιότητα της νομοθεσίας μας. Αυτό διακυδεύεται αυτό και γι' αυτό προτείνω την έσταση και ελπίζω η πλειοψηφία του σώματος να με στηρίξει για να αρχίσουμε πραγματικά με καλύτερη νομοθετική ρύθμιση σήμερα. E Ευχαριστούμε. Να ξεκινήσουμε με τον Πέτερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούστηκε το όνομά μου κατ' επανάληψη και γι' αυτό χαίρομαι που μπορώ να απαντήσω αμέσω. Έχω βέβαια κάποια κατανόηση για την θέση του Μπάς Eichhout και για την θέση των συναδέλφων που υπέβαλαν το σχετικό ψήφισμα. Παρ' όλα αυτά, δυσαρεστούμε πολύ από τη δράση ορισμένων λόμπι. Βλέπουμε λόμπι με ισχυρή επιρροή να αντιδρούν την εμπορία των δικαιωμάτων ε, εκπομπών. Και οι τιμές είναι πολύ χαμηλές τώρα. Έτσι λοιπόν μπορούν απλά να περιμένουμε στα σταυρωμένα χέρια μέχρι ότου το εμπόριο αυτό να πεθάνει ήσυχα. Όμως αμφισβητείται έτσι και ολόκληρη η πολιτική για την προστασία του κλίματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ δεν μπορώ να είμαι σύμφωνος σε αυτό. Εάν τα λόμπι δεν έπαιζαν τόσο άσχημο παιχνίδι τα τελευταία χρόνια και τους τελευταίους μήνες, δεν θα χρειαζόταν καν να κάνουμε τη συζήτηση αυτή. Ο Μπάς Σέικχαουτ μπορεί να είχε τι σχετικέ ενστάσει, αλλά παρόλα αυτά δεν θα έβρισκε τόση μεγάλη απήχηση. Χρειαζόμαστε φιλόδοξη πολιτική από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Φάνηκε καθαρά και στη διάσκεψη κορυφή που οργάνωσε ο Μπάν Κιμούν στην Νέα Υόρκη. Ήταν πραγματικά εξαιρετικά δυσάρεστο που δεν είχε μία ενιαία θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί πρέπει να έχουμε ενιαία θέση ως Ευρωπαϊκή Ένωση. 40% μείωση μέσα στην Ένωση. Αυτό πρέπει να γίνει. Αυτή είναι και η θέση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Δεν τίθεται θέμα για μας για τον αριθμό αυτό που είναι και κρίσιμο διεθνώς. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ενισχύσουμε το εμπόριο των δικαιωμάτων εκπομπών. Γι' αυτό και συμφώνησα με το backloading. Με μεγάλη στήριξη, με ενθουσιώδη στήριξη και του υποψήφιου αρμόδιου επιτρόπου. Είμαι και υπέρ της έκθεσης του Ιβο Βέλετ. Η προσωπική μου γνώμη είναι μάλιστα ότι πρέπει η μείωση αυτή να προταχθεί, να γίνει ήδη από το 2017. Το ότι δεν βρίσκουμε υποστήριξη από τη βιομηχανία, αυτό αποτελεί ένα τμήμα του προβλήματος που οδηγεί στη συζήτηση που διεξάγουμε σήμερα. Εάν ωστόσο προχωρήσει το εμπόριο των δικαιωμάτων εκπομπών δεν θα μιλούμε πλέον για 5 ευρώ, αν είναι σαφές ότι θα εισαχθεί το σύστημα, ότι θα ε, εφαρμοστεί το σύστημα, τότε αποδυναμώνονται και πολλά επιχειρήματα του μπας. Παρ' όλα αυτά είναι δύσκολα τα πράγματα, το δέχομαι. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, τώρα που έχουμε κάνει δύο εντατικές συζητήσεις γι' αυτό, καταλήγουμε ωστόσο να απορρίπτουμε τις προτάσεις του Bas Out. Κάτι που δεν έχετε και ακόμα που όμως είναι κρίσιμο, είναι ότι αυτός ο κατάλογος της διαρροής άνθρακα περιλαμβάνει και επιχειρήσεις που είναι πρωτοπόρες στην τεχνολογία. Μόνο οι 10 πρωτοπόρες τεχνολογικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη λαμβάνουν τα πιστοποιητικά τους δωρεάν. Όλες οι άλλες οφείλουν να συμμετέχουν σε δράσεις και να αγοράζουν τα πιστοποιητικά τους. Μόνο οι 10 καλύτερες λαμβάνουν, το ξαναλέω, τα πιστοποιητικά τους δωρεάν. Εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε την καινοτομία. Θέλουμε να, γίνει, να γίνουν επενδύσεις εδώ στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες που να είναι πραγματικά στην αιχμή της τεχνολογίας και εφόσον το πράξουν αυτό οι επιχειρήσεις δεν θα χρειάζονται πλέον να αγοράσουν πιστοποιητικά για την εκπομπή των, των διοξιδίων ούτε για 5, ούτε για 10, ούτε για 30 ευρώ. Δεν μπορούμε, μπορούμε όμως να τις τιμωρούμε επειδή βρίσκονται, είναι προηγμένες τεχνολογικά. Εμείς θέλουμε να προωθήσουμε την καινοτομία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντική πτυχή του εμπορίου δικαιωμάτων εκπομπών. Και όσες επιχειρήσεις έχουν επενδύσει τα τελευταία χρόνια στις low carbon emissions, τώρα τιμωρούνται με, από την απόρριψη αυτής της λίστας από τη δική μας πλευρά της λίστας, της carbon leak, leaking ε, λίστας δηλαδή. Επαναλαμβάνω ότι αυτό που θέλουμε εμείς είναι μόνο οι προηγμένες επιχειρήσεις. Διατελώς είναι σαν όλες οι ποδοσφαιρικές ομάδες, όπως αν όλες οι ποδοσφαιρικές ομάδες στην Ευρώπη να ήταν πρωταθλητές στην Champions League. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και φέρνω το παράδειγμα και της ε, Bayern με τη Real Madrid. Δεν έφταιγε ο διαιτητής, οι Ισπανοί ήταν καλύτεροι. Έτσι είναι, υπάρχουν καλύτεροι και υπάρχουν και καλοί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει κριτήρια. Όποιος πληρεί τα κριτήρια δεν χρειάζεται να αγοράζει πιστοποιητικά. Και αυτό υποστηρίζει την καινοτομία. Θα είναι λάθος μήνυμα να πούμε στις επιχειρήσεις που θεώρησαν ότι αν κάνουν επενδύσεις θα είναι μεταξύ των πρώτων, να έρθουμε να τους πούμε τώρα, α, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα μετάνιωσε και παρόλα αυτά οφείλει να συμμετάσχεις στο εμπόριο, οφείλει να αγοράσεις τα πιστοποιητικά. Δεν είναι μυστικό άλλωστε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει μια διασύνδεση μέσα στις εσωτερικές της συζητήσεις. Τα 40%, τα 40 μείωση που θέλουμε και που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι συμφώνησε γιατί υπήρχαν και επίτροποι που δεν ήθελαν το 40% μείωση. Και τώρα μία μέρα μετά από τη διάσκεψη κορυφής του Μπαν Κιμούν πρέπει να τα δούμε τα πράγματα. Τώρα πας εσύ λες ότι δεν θέλεις να ανατρέψεις ολόκληρο τον κατάλογο, ολόκληρη τη λίστα. Θες να την αλλάξεις, όμως αυτό νομικά δεν γίνεται. Σήμερα το ερώτημα που τίθεται είναι ναι ή όχι. Νομικά έχουμε ένσταση που επιτρέπει να απορρίψουμε ολόκληρη τη λίστα. Μπορούμε να πούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κοιτάξτε θέλουμε άλλη λίστα, αλλά ποια θα είναι η μορφή τη άλλη λίστας δεν είναι γραμμένο πουθενά, γι' αυτό νομικά έχουμε μόνο το δικαίωμα να πούμε ναι ή όχι. Άρα αυτό που λέμε είναι ότι εφόσον προβάλλουμε ένσταση, απορρίπτουμε τη λίστα. Αυτό σημαίνει όμως πάλι ότι καμιά επιχείρηση σε κανένα κλάδο της οικονομίας δεν θα έχει ασφάλεια για το μέλλον. ομολογώ και το είπα και από την αρχή ότι εδώ υπάρχουν πολλοί που είναι υπεύθυνοι και υπάρχει και λάθος στάση πολλών λόμπι εδώ στις Βρυξέλλες. Αυτό όμως δεν επιτρέπεται να αποβεί τελικά σε βάρος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που ωστόσο αυτές θα την πληρώσουν εάν υποστηρίξουμε σήμερα την ένσταση. Γι' αυτό τελικά το Λαϊκό Κόμμα τίθεται αντίθετο με την ένσταση του Μπρας Eichhout. Σας ευχαριστούμε κύριε Λίζα. Κύριος Γκρότερ. Η δική μας η πολιτική ομάδα, λέει ο Ματίας Κρότε των Σοσιαλιστών, δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη. Αναμένουμε τη σημερινή συζήτηση που θα διεξαχθεί και με την Κομισιόν. Εγώ προσωπικά έχω μεγάλη κατανόηση για την ένσταση του Bass Eichhout, διότι τελευταία ασχοληθήκαμε πολύ με αυτό το λεγόμενο backloading για το πώς θα προωθήσουμε και πάλι το εμπόριο των δικαιωμάτων ε, εκπομπών. Έχουμε και την έκθεση του Ιβο για μια σταθεροποίηση της αγοράς, έτσι ώστε το εμπόριο των πιστοποιητικών να μπορέσει να αναπνεύσει, να μπορεί να παρακολουθήσει και τις ε, διακυμάνσεις της συγκυρίας, της οικονομικής συγκυρίας. Κανείς δεν είναι τρελός να πει ότι απορρίπτω απολύτως την Carbon Leaking List και επομένως να σηκωθούν να φύγουν όλες οι επιχειρήσεις από την Ευρώπη. Κανείς το θέλει αυτό. Όμως το ανακοινωθέν τύπου του Λίζε κάπως έτσι παρουσιάζονταν τα πράγματα. Και αυτό είναι παραπλανητικό για την κοινή γνώμη. Από τη μια μεριά ακούμε ωραίους λόγους, στην διάσκεψη κορυφής του Πανκιμούν πάνε οι Ευρωπαίοι, λένε ωραία πράγματα. Όταν όμως έρχεται ο κόπος το χταίνει, τότε λένε «Α, θα προχωρήσουμε, αλλά με τραβηγμένο το χειρόφρενο». Θυμίζω τις συζητήσεις για το backloading, γιατί για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό το θέμα και πραγματικά ε, άσπεσαν τα μαλλιά μου σε ένα βαθμό από αυτή την ιστορία. Έχουμε πολλά πιστοποιητικά στην αγορά, υπερβολικά πολλά. Γι' αυτό και λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιε θα είναι οι επιπτώσεις αν λάβουμε ως βάση τα 30 ευρώ τον τόνο ή τα 16 ευρώ τον τόνο. Αυτά θέλω να τα ξανακούσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι σημαίνει αυτό για την ποσότητα των πιστοποιητικών εάν δεχθούμε την ένσταση του ΕΚΑ ότι αν την απορρίψουμε. Τι σημαίνει αυτό και για τον τελικό λογαριασμό. Για την ώρα η τιμή είναι στα 5 ευρώ τον τόνο. Και εσείς μιλάτε για 30 ευρώ τον τόνο. Υπάρχει μια διαφορά 25 ευρώ. Ποιος την πληρώνει τη διαφορά αυτή. Τη διαφορά την πληρώνουν οι απλοί πελάτες των επιχειρήσεων ενέργειας. Για εξηγήστε μας λίγο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τελικά ποιος θα αναγκαστεί να πληρώσει για τα πλεονεκτήματα αυτά υπέρ της βιομηχανίας. Και τέλος, αν δεχθούμε σήμερα την πρόταση του Μπάς Eichhout, να υπερψηφίσουμε δηλαδή, τι σημαίνει στην περαιτέρω πορεία. Αν τα γνωρίζω καλά, μέχρι τον Απρίλιο του 2016 θα πρέπει να αγοράσουν πιστοποιητικά οι ε, επιχειρήσεις. Βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρεί αργά, αδιαφανώς κάνει μελέτη που την οποία δεν καθιστά ακόμα δημόσια, έτσι διαμορφώνεται εδώ μια τάση του Κοινοβούλου να απορρίψει. Και εφόσον γίνει δεκτή η carbon leaking λίστα, θα πρέπει να γίνει αυτό μέσα σε 4-5 μήνες. Γι' αυτό θέλω να γνωρίζω ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στον αριθμό των πιστοποιητικών. Αυτό που είπε για τα λόμπι ο Πετρελίζη είναι σωστό, ωστόσο. Ορισμένοι προσπάθησαν να εμποδίσουν το backloading. Είπαν ότι 5, 5 δολάρια μάλλον τον τόνο είναι υπερβολικά πολλά ούτως ή άλλως. Θα έπρεπε να, η, η πραγματικότητα θα έπρεπε να είναι να μειώσουμε την τιμή στα 5 ευρώ. Κανένα δεν θέλει ωστόσο να θάψει την λίστα του carbon leakage. Αλλά ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο. Θα πρέπει να προσαρμοστεί η λίστα στην πραγματικότητα. Διότι κάποια στιγμή ο κόσμος έξω θα πάψει να δέχεται πλέον την ανάγκη προστασίας του κλίματος και κυρίως το ότι πρέπει να πληρώνει για την προστασία του κλίματος. Δεν μπορεί ένα μέρος να απαλλάσσεται, ένα τμήμα της οικονομίας να απαλλάσσεται και ένα άλλο να επιβαρύνεται για να έχει τα προνόμια το πρώτο μέρος. Αυτές είναι οι ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πολιτική μου ομάδα θα επανέλθει στο θέμα αυτό σήμερα για να το συζητήσει. Δεν είναι βέβαια απλό το θέμα, δεν μπορεί κανείς να το λύσει αυτοσχεδιάζοντας. Επαναλαμβάνω ότι τα λόμπι φέρουν βαριά ευθύνη. Θα μπορούσα να ονοματίσω και ορισμένα, αλλά προτιμώ να τα αφήσω για σήμερα. Ευχαριστούμε ο κύριος Ντάνκαν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευθύ εξ αρχή να πω ότι συμφωνώ με τον κύριο Έικχαουτ για τη μελέτη αντικτύπου θα έπρεπε να την έχει σεβαστεί η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπήρχε χρόνο γι' αυτό. Όμω, εμεί ω ομάδα δεν θα στηρίξουμε την ένστασή του. Πρέπει να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε και είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω είναι γνωστό σε όλου ότι το σύστημα ανταλλαγή και εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών δεν λειτουργεί όπω θέλαμε. Νομίζω ότι όλοι το ξέρουμε. Έχει εντωμεταξύ όμω από τότε που ξεκίνησε να χρησιμοποιείται το σύστημα, επέλθει και η οικονομική κρίση, η οποία έχει τεράστιε συνέπειε για τον κλάδο αυτό και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Και ήδη έχουν αλλάξει τα επίπεδα δραστηριότητα του βιομηχανικού τομέα. Θα πρέπει λοιπόν το θέμα της διαρροής του άνθρακα να το βλέπουμε και στο πλαίσιο αυτό της οικονομικής κρίσης. Το σύστημα αυτό ανταλλαγής αυξάνει την τιμή ε, των εκπομπών του άνθρακα. Κάτι που ε, πίεζε, για το οποίο πίεζε το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας, δηλαδή να υπάρχει backloading και να, υπά, να είναι η τιμή ψηλά στα 30 ευρώ ανά τόνο. Αυτό αναγνωρίζεται από όλους. Νομίζω όμως ότι σε αυτή την συγκυρία αντιμετωπίζουμε μια πρόκληση. Να δούμε την έσταση αυτή και αν θα τη στηρίξουμε ή όχι. Εάν τη στηρίξουμε θα δημιουργήσουμε ένα πρόβλημα. Δεν είναι θέμα απλής απόφασης βεβαίως, είναι μια διτή απόφαση. Εάν στηρίξουμε την ένσταση, δημιουργούμε στάθειες σε εταιρείε και βιομηχανίε, οι οποίε αυτή τη στιγμή χρειάζονται το αντίθετο. Θα πρέπει, εφόσον αυτό φτάσει στον Ιλομελία, να φτάσουμε σε υλοποίηση των όσων θα ορίζει η ένσταση με ένδικα μέσα και να δούμε τι συνέχεια θα δώσουμε στην ένσταση. Εάν δεν έχουμε ένα κατάλογο για το 2015, θα έχουμε σημαντική αστάθεια και θα δημιουργήσουμε νομικό κενό. Νομικό κενό για τι εταιρείε τι οποίε αφορά η ένσταση. Αυτό πιστεύω θα ήταν πρόβλημα. Ο στόχο μα είναι να προσφέρουμε σταθερότητα στην ε, βιομηχανία και το σχετικό βιομηχανικό κλάδο για να μπορέσει να υπάρξει ανάκαμψη. Το σώμα μα θέλει ένα σύστημα ανταλλαγή, ένα σύστημα εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών που να λειτουργεί. Νομίζω υπάρχουν πολλέ άλλε μέθοδοι για να το επιδιώξουμε ως στόχο κάτι τέτοιο. Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους νομίζω δεν πρέπει να στηρίξουμε την ένσταση και γι' αυτό η ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών δεν θα υπερψηφίσει την ένσταση. Ευχαριστώ. Okay, Mr. Ευχαριστούμε κύριος Γκυρμπράντη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θεωρώ ότι μεγάλο μέρος της πλειοψηφίας όσων παρόντα την αίθουσα είναι υπέρ τη Ευρωπαϊκή Ένωση όπω και εγώ ίδιο. Εμεί, οι υπέρμαχοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση, περάσαμε μια πολύ δύσκολη προεκλογική εκστατεία. Με ένα, με ένα εκλογικό σώμα που όλο ένα και περισσότερο επικρίνει την χάραξη πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ ε, είμαι υπέρμαχος της ε, διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε σχέση με το εθνικό επίπεδο. Θεωρώ ότι οι ευρωπαϊκές αποφάσει είναι πολύ πιο διαφανεί και μάλιστα στη διαδικασία λήψη αποφάσεων από ότι στις, στα εθνικά κράτη. Αλλά πρέπει να επικεντρωθούμε και στου μακροπρόθεσμου στόχου μα. Την ίδια στιγμή που το Εθνικό μα Κοινοβούλιο είχε μια μακροσκελέστατη συζήτηση για κάτι που συνέβαινε στην Βόρεια Ιλλανδία, εμεί συζητούσαμε την ενεργειακή μα κατάσταση ω το 2050. Είναι και θέμα μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση. Ε, η ευρωπαϊκή λήψη αποφάσεων είναι πιο σημαντική από, την εθνική, από τις εθνικές αποφάσεις, διότι ακριβώ βασιζόμαστε και σε επιστημονικά στοιχεία, σε μελέτες αντικτύπου που δημοσιεύονται. Την πολιτική μας και τη χάραξή της τη βασίζουμε σε μελέτες αντικτύπου. Είναι λοιπόν συνήθως ε, πολύ ενδελεχείς και πολύ καλά τεκμηριωμένες οι αποφάσεις μας. Και τώρα φτάνουμε στην πρόταση για τη διαρροή του άνθρακα η οποία βασίζεται σε μια αδημοσίευτη μελέτη αντικτύπου και μάλιστα αντιφάσκοντας με αυτή την αδημοσίευτη μελέτη. Η πρώτη μου ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν είναι γιατί φτάνουμε να έχουμε αυτή τη συζήτηση χωρίς δημοσιευμένη μελέτη αντικτύπου. Και από πού και ως πού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντάσσει πρόταση που δεν συνάδει με την δική της την μελέτη, την ίδια όχι απλώς αποκλίνει λίγο από την δική της μελέτη, αλλά είναι τελείως αντίθετη. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει κάποια εξήγηση. Εάν λαμβάνουμε σοβαρά ε, την υπόψη, εάν παίρνουμε στα σοβαρά μάλλον την ε, χάραξη πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και ω προ τι ευρωπαϊκέ εταιρείε, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε μακροπρόθεσμη και επιστημονικά τεκμηριωμένη και αποτελεσματική και διαφανή ε, προσέγγιση. Τα 30 ευρώ ανά ε, δεν έχουν καμία σχέση με όσα τα επιστημονικά στοιχεία σε αυτό το τομέα μας ε, μαρτυρούν. Να τονίσω λοιπόν αυτό που είπε και ο Μπάς, ότι η ίδια διαρροή του άνθρακα δεν είναι ακριβώς το αντικείμενο της συζήτηση, αλλά είναι ο τρόπος που υπολογίσαμε, που υπολογίσαμε και διατυπώσαμε και συντάξαμε αυτόν τον κατάλογο. Το σύστημα εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών, η διαρροή του άνθρακα, οτιδήποτε μα επιτρέπει να καταπολεμήσουμε τι αλλαγέ του κλίματο, βασίζεται στην υπόθεση ότι θέλουμε να τονώσουμε την καινοτομία. Εάν θέλουμε να τονώσουμε την καινοτομία, Πρέπει να ε, συνδράμουμε τις εταιρείες οι οποίες όντως επενδύουν στην καινοτομία. Θα πρέπει λοιπόν να επιδιώξουμε, να τις εξωθήσουμε ή μάλλον να εξωθήσουμε τις εταιρείες που δεν επενδύουν στην καινοτομία να το κάνουν. Με αυτό όμως τον κατάλογο της έκθεσης των κίνδυνων διαρροής άνθρακα δεν τις, ε, ε, δεν τις παροτρύνουμε να κάνουν κάτι τέτοιο ούτε θα επιδιώξουν οι εταιρείε αυτές να επενδύσουν στην καινοτομία. Νομίζω η ψηφοφορία αυτή είναι μια ψηφοφορία απόλυτη όπου θα πρέπει να πούμε ναι ή όχι στο αντικείμενο της ψηφοφορίας. Εάν όμως πούμε όχι στον κατάλογο διαρροής του άνθρακα δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει κανένας κατάλογος στο μέλλον. Μπορούμε να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντάξει ένα καλύτερο κατάλογο μεταγενέστερα. Και ως ε, από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές χαίρομαι πολύ που ακούω ότι θέλουν και οι συντηρητικοί μεταρρυθμιστέ να ανέβει η τιμή του άντρακα στα 30 ευρώ ανά τόνο. Χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ που ακούω αυτή την υπόσχεση από του συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ και με τα χαρά να συνεργαστούμε μαζί σα όταν θα δούμε τι διορθώσει στο σύστημα εμπορία δικαιωμάτων του ερχόμενου μήνε. Αναμένω λοιπόν τι προτάσει σα και τη στήριξή σα. Ε, ε εν τέλει Κύριε Πρόεδρε, χθε οργανώθηκε η Σύνοδο Κορυφή για το Κλίμα στην Νέα Υόρκη. Και είδαμε τι πρώτε ειδήσει από τη Σύνοδο αυτή. Δηλώσει ότι η ιδέα μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη εμπορίας ε, και η εξισορρόπηση αλλαγών του κλίματος και αγοράς είναι μια λανθασμένη προσέγγιση, ακόμη και αν δούμε τα πράγματα μονομένα αναγεωγραφική ζώνη δεν σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίσουμε το και στο κλίμα, καταστρέφουμε την οικονομία μας. Αν χρησιμοποιήσουμε το σύστημα εμπορία, ε, κάνουμε πιο ισχυρή την οικονομία μα. Και αυτό δεν το λένε οι μη κυβερνητικέ οργανώσει, αλλά ε, το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και η Διεθνή Επιτροπή για το Κλίμα, όπου πολλοί σεβαστοί και επαείοντε έχουν εργαστεί για να καταλήξουν σε αυτά τα συμπεράσματα. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν θα υπερψηφίσω την ένσταση και πραγματικά σπιέσουμε πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, να καταρτήσει ένα νέο κατάλογο διαρροής του άνθρακα που να βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία και όχι σε εμπορικέ συμφωνίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. κυρία Ευχαριστώ πρόεδρε. Ως ε, ομάδα θα υπερψηφίσουμε την ένσταση. Θέλουμε να στείλουμε ένα περισσότερο πολιτικό και κοινωνικό μήνυμα, ίσως και λιγότερο τεχνικό. Αντιλαμβανόμαστε ως ομάδα ότι το θέμα της εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών <clears throat> έχει καταλήξει να αποφέρει μεγάλο κέρδος στις μεγάλες επιχειρήσεις που ρηπαίνουν περισσότερο. Πρώτα απ' όλα έτσι δίνονται δωρεάν τέτοια δικαιώματα. Αυξάνοντας την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος που πληρώνει ο καταναλωτής, πρώτα απ' όλα, ενώ θα μπορούσε να μην συμβαίνει αυτό. Και έπειτα κερδοσκοπούνε με τις ποσοστώσεις εμπορίες δικαιωμάτων ε, εκπομπών. 2015 με 2020 θα έπρεπε να γίνει η κατανομή λοιπόν των δωρεάν αυτών δικαιωμάτων. Αλλά η βιομηχανία πίεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρει ένα άλλο άλοθη για να δώσει δωρεάν τέτοια δικαιώματα. Ο κατάλογος που έχουμε μπροστά μας καταλήγει να μπορεί να αποφασίσει μία βιομηχανία αν της επιβληθεί κάποιο ποσό να απειλεί με το ότι θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα είναι εκβιασμός αυτός. Δεν είναι σωστό όμως να γίνεται ένας τέτοιος εκβιασμός. Έπειτα, ο υπολογισμός, όπως ακούσαμε, βασίζεται όχι σε αντικειμενικά δεδομένα, αλλά σε ένα υποθετικό ποσό. 30 ευρώ ο τόνος του οξύδιου του άνθρακα, ενώ ξέρουμε ότι σήμερα είναι 5. Το πολύ 5. Ο κίνδυνος μετακατάστασης όμως δεν δικαιολογείται κατά τη γνώμη μας. Πρόκειται για ένα άλοθη απλώς και μόνο. Γι' αυτό και στηρίζουμε την ένσταση, γιατί δεν θέλει να συνεχίζουμε να επιδοτούμε ρηπαίνουσες βιομηχανίες. Είμαστε κατά εξάλλου του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, γιατί το αποτέλεσμα είναι το κέρδος της βιομηχανίας και τίποτα άλλο. Και δεν μειώνονται τελικά οι εκπομπές στην πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Πίτερ Λίζε εξέφρασε πολύ καλά την θέση της ομάδας μας. Θέλω όμως να υπογραμμίσω ότι το θέμα της βεβαιότητας στο σχεδιασμό είναι ένα πολύ σημαντικό επιχείρημα και υπενθυμίζω ότι το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών όπως θα έχει από 1η Ιανουαρίου 2015 Ισχύει δηλαδή μετά από λίγες εβδομάδες, λίγους μήνες. Δεν είναι μόνο πολιτικό το ζήτημα όμως, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις τεχνικές προδιαγραφές. Μπορούμε να απαντήσουμε με ναι ή με όχι από ό,τι φαίνεται. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καταρτήσει νέο κατάλογο αν πούμε όχι. Με όλες τις καθυστερήσεις και τις δυσκολίες. Συνεπώς, είναι και θέμα χρονοδιαγράμματος. Πρέπει να δράσουμε και να μην υποστηρίξουμε την ένσταση. Ευχαριστώ, παρακαλώ. Η κυρία Γκροστέτ, πρόεδρε, δεν άκουσα καθόλου το όνομά μου. Ο Πέτερ Λίζε πολύ σωστά ανέπτυξε τη θέση της ομάδας μας, του ΕΛΚ, και στηρίζω απολύτως την τοποθέτησή του. Νομίζω ότι η απόρριψη του καταλόγου των τομέων, διότι για καταψήφιση μιλάμε ουσιαστικά, των ε, τομέων που εκτίθενται στη διάρκεια του άνθρακα θα δημιουργούσε αβεβαιότητα. Αβεβαιότητα την οποία δεν χρειάζονται οι επιχειρήσεις ως προς την προβλεψιμότητα για τις επενδύσεις τους. Σε ένα πλαίσιο οικονομικής κρίσης και αύξηση των τιμών της ενέργειας, οι ευρωπαϊκές εταιρείες χρειάζονται στήριξη. Χρειάζονται στήριξη για να αντιμετωπίσουν την ε, διεθνή ανταγωνισμό και να υπάρξει βιομηχανική άνθηση στην Ευρώπη. Χρειάζονται σταθερότητα. Η τιμή του άνθρακα που χρησιμοποιείται ω τιμή αναφορά για να καθοριστούν οι τομεί που είναι εκτεθειμένοι στον κίνδυνο διαρροή δεν είναι επαρκώ δικαιολογημένη. Να θυμίσω ότι ένα τομέα δράση στην στον κατάλογο αυτό δεν σημαίνει ότι απαλλάσσεται από τις ευθύνες για μείωση των εκπομπών ίσα ίσα με τους άλλους τομείς του συστήματος ε, του, των ανταλλαγών δικαιωμάτων εκπομπών από το 2005 στο 2020 πρέπει να κάνει την προσπάθεια μείωσης κατά 21%. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι κάποιες επιχειρήσεις δικαιούνται την ότι δεν δικαιούνται όλες οι επιχειρήσεις της ποσοστώσεις 100% δωρεάν αλλά μόνο αυτές που βάσει του benchmarking έχουν εγκαταστάσεις ε, οι οποίες επιτρέπουν να μην υπάρχει διαρροή του άνθρακα αυτές θα λάβουν μόνο και αυτές τις υποδομές και για το υπόλοιπο των εγκαταστάσεών τους θα πρέπει να δίνουν τις σχετικές προσπάθειες. Οι επιχειρήσεις λοιπόν που έχουν δωρεάν ποσοστώσεις δεν θα έχουν τέτοιες, ε, τέτοια ωφέλη στην περίπτωση που ο διορθωτικός παράγοντας ε, διατομιακός εφαρμόζεται ετησίως άνω του 17% για το 2020 θα λάβουν μόνο όσες ε, έχουν συγκεκριμένες υποδομές που επιτρέπουν την ε, μη ε, εκπομπή άρθρακα. Εδώ λοιπόν πρέπει να λαμβάνουμε πόσο και την οικονομική προτεραιότητα πέρα από τις περιβαλλοντικές μας μερίμνες και να μην ξεχνάμε ότι η πραγματικότητα αυτή είναι πολύ σκληρή στην Ευρώπη και όλε τι εταιρείε. Αυτό ήθελα να πω για να στηρίξω τη θέση του ΕΛΚ. Ευχαριστούμε η συνάδελφος Γκούτλαντ. Ευχαριστώ. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και αξίζει το θέμα βέβαια να εμβαθύνουμε περισσότερο. Η πρόταση του Μπάς Εκχούτ είναι πολύ ενδιαφέρουσα και μπορεί να αποτελέσει μια πάρα πολύ καλή βάση για να ξεκινήσουμε από αυτήν. Βλέπω ότι ξεκάθαρα υπάρχουν επιχειρήματα για να αφισβητήσουμε τα κριτήρια τα οποία στηρίζουν την κατάρτιση του καταλόγου αυτού, όπως η τιμή. Όπως είπανε πολλοί, οι τιμές είναι πολύ χαμηλότερες ανατόνο τόνο διοξιδίου του άνθρακα. Βασίζεται η Επιτροπή στα 30 ευρώ. Μα νομίζω ότι αυτό είναι και η καρδιά της συζήτησης ουσιαστικά. Οι συνέπειες από τον υπολογισμό αυτών. 16% θα έπρεπε να ήταν ο υπολογισμός να βασίστε το 16% και όχι στην τιμή των 30%. Άρα πρέπει να πάει πίσω η πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να μας προτείνει κάτι νέο που να βασίζεται στον υπολογισμό βάσει πιο ρεαλιστικής τιμής. Πρέπει Σήμερα λοιπόν να έχουμε υπόψη μας ότι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνε μας. Με ένα σύστημα το οποίο τελικά να μειώνει την ρήπανση και τις εκπομπές του του άνθρακα. Νομίζω ότι η... τόσα λέει το ΕΛΚ δεν είναι τόσο προδευτικά προκειμένου να μειωθεί η ρήπανση στην Ευρώπη. Εμείς νιώθουμε την ευθύνη Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να υπάρχουν επενδύσεις πράσινες που να βοηθήσουν την Ευρώπη να πάει μπροστά στο θέμα του περιβάλλοντος. Η επιχειρηματολογία του ΕΛΚ. Μου φαίνεται σαν να λέγαμε σε έναν έφηβο δεν χρειάζεται να διαβάσει τώρα τα μαθήματά σου και να προετοιμαστεί για εξετάσει, για το θέμα που θα σου πέσει αύριο μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που διαβάζει. Φρόντε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτές τις μέρες, όταν μάθαμε ότι θα συζητηθεί το θέμα αυτό, πρέπει να πω ότι δεχτήκαμε φοβέρε πιέσεις από τις ομάδες συμφερόντων, οι οποίοι δεν ε, δίστασαν καθόλου να μας στείλουν τις απόψεις τους και το ποιε είναι οι προτεραιότητέ του. Όμω, εμεί ω κίνημα Τσίνκου Εστέλε έχουμε πολύ καλέ σχέσει με του πολίτε και μαθαίνουμε και εκείνοι τι γνωρίζουν και τι πιστεύουν. Μα έγραψαν και εκείνοι λοιπόν από την πλευρά του σχόλια ε, για... και ερωτήσει για το πώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εφαρμόσει σωστά ε, μια από τι θεμελιώδει αρχέ τη συνθήκη ε, τη Λισαβόνα. Η... Τη ε, αναχέτηση τη ρήπανση. Η το πώς θα λάβει υπόψη στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση το λόγο των πολιτών. Πώς επιτρέπει επίση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 50% των εταιριών που είναι πλέον υπογόνες να έχουν μηδενικέ ποσοστώσεις. Ή πώς μπορεί το σύστημα εμπορία δικαιωμάτων των εκπομπών να συμφωνεί με το στόχο ε, να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα 90% στο 2050. Πώς ε, μπορεί να θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το σύστημα αυτό ε, εμπορίας θα μας φέρει τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα τα οποία έχει πει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι επιδιώκει. Εμείς λοιπόν ως κίνημα στόχο έχουμε να ε, φέρουμε εδώ τη φωνή των πολιτών. Μας ζητούν λοιπόν να στηρίξουμε την ένσταση του συναδέλφου και να καταργήσουμε τον κατάλογο αυτό. Ως ε, ομάδα EFD λοιπόν θα υπερψηφίσουμε την ένσταση. Η κυρία Κονέτσινα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, η δική μου φωνή θα διαφέρει λίγο από τις παρεμβάσεις των άλλων συναδέλφων. Η δική μου χώρα έχει μεγάλο ποσοστό βιομηχανίας έντασης ενέργειας. Το μόνο που ζητώ εγώ είναι μια λογική στάση. Αν είχαμε κάνει τις προτάσεις αυτές προεξαμήνου, θα ήταν κατανοητό, διότι θα είχαμε χρόνο να τις συζητήσουμε. Τώρα όμως βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου αν πούμε ναι στην ένσταση Eichhout, καταλήγουμε σε μια αβεβαιότητα, σε μεγάλο αριθμό κλάδων της βιομηχανίας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Μιλούμε σήμερα για αύξηση της ανεργίας που δεν μπορούμε πια να αντιμετωπίσουμε. Μπορεί να συμβεί οπουδήποτε αυτό. Θα καταλήξουμε σε σοβαρό πρόβλημα που οφείλουμε να το αναμένουμε. Πρώτη προτεραιότητα για μας θα πρέπει να είναι η σύγκριση και εξισορρόπηση όλων των πτυχών του περιβάλλοντος και μια εναρμόνιση μεταξύ τους. Για μένα λοιπόν είναι απαράδεκτο να οδηγήσουμε τα θεσμικά όργανα σε μια νομοθετική παγίδα. Το γεγονός ότι την πρόταση της Επιτροπής την υποστηρίζουν 27 χώρες μέλη είναι μια ένδειξη. Το όλο θέμα έχει συζητηθεί σε βάθος και το έχουν υποστηρίξει, τις προτάσεις αυτές έχουν υποστηρίξει και οι εθνικοί εμπειρογνώμονε. Εγώ θα ήθελα να δω μελέτη αντικτύπου για τις επιμέρους χώρες. Για τη δική μου χώρα, την τσεχική δημοκρατία δηλαδή, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο. Ευχαριστούμε Αντιπρόεδρο Σποτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πραγματικά η συζήτηση είναι αρκετά απογοητευτική. Φαίνεται να βρισκόμαστε σε πίεση. Εάν ακούω ότι τα λόγια της συναδέλφου της ΓΚΟΕ από την ε, Τσεχική Δημοκρατία, βρισκόμαστε σε πίεση. Όλοι μας πιέζουν. Οι λομπίστες, οι μηχανίες, οι εταιρείε. Καλούμαστε να αναλάβουμε ευθύνες και ούτω καθεξής. Ναι, έτσι είναι. Συζητούμε ένα τεχνικό θέμα και προσπαθούμε να είμαστε συνετοί. Αυτό είναι σαφές. Αλλά υπάρχουν δύο ζητήματα πολύ σοβαρά. Το πρώτο είναι γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσέβεται την ίδια της τη μελέτη αντικτύπου. Και ποια είναι τότε η αξία μιας τέτοιας μελέτης. Ποια είναι η αξία της λήψης ε, ...της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ίδια δεσέβεται τη δική της τη μελέτη. Αυτό λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε να ακουστεί. Και το δεύτερο κατά την άποψή μου είναι ότι εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων δημιουργεί συνέπεια, ε, προκαλεί ασυνέπεια. Εμείς πρέπει να το, να το δεχτούμε αυτό και να το ε, συνεχίσουμε, να επιτρέψουμε να συνεχίζεται. Νομίζω πως όχι. Όπως είπε ο ε, Ματίας, θα το συζητήσουμε στους σοσιαλιστές και δημοκράτες και θα δούμε τι απόφαση θα Αλλά δεν νομίζω ότι η συζήτηση πρέπει να πάψει εδώ και αργότερα ασχέτως της συγκεκριμένη απόφασης για την ένσταση, υπέρ ή κατά, αν θα στηρίξουμε ή όχι την ένσταση, Ασχέτως αυτού θα πρέπει να συζητήσουμε πώς είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μισεύεται την ίδια της τη μελέτη. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Πρόεδρε Πότ. Η συνάδελφος Μπόιλαμ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον Μπάς για την πρότασή του. Νομίζω ότι πρέπει πραγματικά να απορρίψουμε τον κατάλογο, να καταψηφίσουμε τον κατάλογο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι εταιρείε που είναι εκτεθειμένε στον κίνδυνο διαρροή του άνθρακα. Νομίζω ότι η εμπιστοσύνη του κοινού στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρύβει τα αποτελέσματα τη ίδια τη μελετή αντικτύπου τη και αυτό σημαίνει ότι εφόσον μιλάμε για καινοτομία, ε, ε, φαίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενδιαφέρεται μόνο στους, στην αριθμητική καινοτομία. Ε, η τιμή 30 ευρώ ανατόνο είναι ουσιαστικά πάρα πολύ ψηλή. Και η οι μηδενικέ ποσοστώσει που δίνονται σε κάποιε εταιρείε ουσιαστικά ε, είναι, είναι διασπάθηση των ε, χρημάτων των φορολογουμένων και όχι κάτι το δίκαιο. Έτσι λοιπόν το ΣΕΔΕ είναι ένα σύστημα γεμάτο ε, ελαττώματα. Και δεν έχει καμία ε, καλή εικόνα προς το κοινό. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη του κοινού εδώ. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι θέλει να μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, όχι να στηρίξει τις μεγάλες βιομηχανίες που μπορούν να πληρώνουν για να ρηπαίνουν όσο τους χρειάζεται. Ευχαριστούμε. Η συναδελφός Γκαρθία Περέφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι παρεμβάσεις που ακούσαμε μέχρι τώρα από τις διάφορες ομάδες δείχνουν πόσο περίπλοκο είναι αυτό το ζήτημα. Και είναι αλήθεια ότι έχει και ένα τεχνικό σκέλος πολύ σημαντικό, αλλά τελικά μιλάμε πιο πολύ για πολιτικές αποφάσεις. Υπάρχει το τεχνικό ζήτημα, υπάρχει όμως και το πολιτικό ζήτημα, γιατί η απόφαση που θα πάρουμε εδώ ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή, ως ε, Κοινοβούλιο, παρόλο που το θέμα είναι και τεχνικό, θα επηρεάσει διάφορους κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες. Συνεπώς πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πόσο σύνθετο είναι το ζήτημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρέπει να έχει καμιά αμφιβολία ότι θεωρούμε πολύ χρήσιμο τον κατάλογο αυτό για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Όμως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ώστε το σύστημα να είναι επαρκώς ευέλικτο. Δεν πρέπει να υπάρχουν στρεβλώσεις εξαιτίας ε, λανθασμένων τιμών ανατόνο διοξιδίου του άνθρακα. Αν υπάρχει μια σωστή τιμή ως κριτήριο για να καθορίσουμε τις εταιρείε που θα εξαιρούνται ή όχι, αυτό έχει φυσικά πλεονεκτήματα. Συγχρόνως θέλουμε και σταθερότητα στην αγορά. Όμως τα κριτήρια που προτείνει πρόταση τροποποιεί τελικά τον κατάλογο των κλάδων και των επιχειρήσεων και αφήνει απ' έξω κάποιες ε, επιχειρήσεις οι οποίες υπολόγιζαν με τα 30 ευρώ να είναι μέσα στον κατάλογο. Γι' αυτό λέω ότι ανάλογα με την απόφαση που θα πάρουμε θα αλλάξει η πραγματικότητα για ορισμένες επιχειρήσεις που έχουν κάνει τις προβλέψεις τους, τον προγραμματισμό τους. Γι' αυτό πρέπει να ζυγίσουμε τις επιπτώσεις. Είμαι υπέρ του να χρησιμοποιηθεί σαν κριτήριο μια σωστή τιμή διοξιδίου του άνθρακα, αλλά να έχουμε και ένα σύστημα ευέλικτο το οποίο να βοηθάει να καλυφθούν οι δυναμίες του παρελθόντος. Κινδυνεύουμε να πλήξουμε την βιομηχανία, αν αλλάξουμε τον κατάλογο, ότι μας αρέσει είτε όχι τη βιομηχανία, η οποία είναι σημαντική για τόσους πολίτες. Γι' αυτό εκφράζω τις αμφιβολίες μας και όπως είπε και ο συνάδελφος και συντονιστής των σοσιαλιστών, ο κύριος Γρότε, θα το συζητήσουμε παρετέρω στην ομάδα μας για να αποφασίσουμε τελικά. Τη στάση θα κρατήσουμε δηλαδή. Ευχαριστούμε. Ολοκληρώσαμε με τις παρεμβάσεις των ε, συναδελφών. Δεν νομίζω ότι ξέχασα κανένα. Και τώρα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο κ. Μπέγκμαν. Για να απαντήσει σε μια σειρά από ερωτήσεις που τέθηκαν από τους συναδέλφους. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που με επιτρέπετε να κάνω κάποια σχόλια. Πρόκειται για ένα θέμα πολύ σοβαρό. Και να πω ότι η σχετική οδηγία για το ΣΕΔΕ προβλέπεται ο κατάλογος να εγκριθεί μετά από συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όταν λοιπόν έγινε η πρόβλεψη αυτή στην οδηγία, ήταν ήδη γνωστό ότι για τον σχετικό βιομηχανικό κλάδο το θέμα είναι πολύ σημαντικό και ότι θα έπρεπε να ληφθεί απόφαση. Ένα πρώτο σχόλιο για τη μελέτη αντικτύπου. Πράγματι, εκπονήθηκε μελέτη αντικτύπου ήταν γνωστή στα κράτη-μέλη όταν συζήτησαν το σχετικό θέμα. Τα κράτη-μέλη λοιπόν ψήφισαν και συμφώνησαν σχεδόν ομόφωνα, με μόνο μία αποχή, να ληφθεί το μέτρο αυτό. Επίσης, διατέθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο και τα μέλη του. Οπότε δεν είχαμε καμία πρόθεση να αποκρύψουμε κάτι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε από τους ε, βουλευτέ. Απλώ ήταν Προφανώ προφανώς ήταν απαραίτητο να αξιολογηθεί το σχέδιο αυτοπόφαση. Βεβαίω υπάρχουν πολλά οικονομικά και πολιτικά επιχειρήματα, αλλά σε αυτή την ε, μελέτη αντικτύπου προβλέπεται υποχρέωση από την οδηγία ΦΕΔΕ να να συνταχθεί ο κατάλογο και αποφασίσαμε απλώ να ακολουθήσουμε αυτή την ε, υποχρέωση. Πρώτα απ' όλα υπήρχαν πολλά νέα δεδομένα λέει και η οδηγία ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα από την τελευταία τριετία. Χρησιμοποιήσαμε λοιπόν στοιχεία για τι εκπομπέ, για την κατανάλωση ηλεκτρισμού, για την κίνηση τη βιομηχανία και ούτω καθεξής. Τα βασικά τώρα σημεία για να είναι κανεί στον κατάλογο πρέπει να ξεπερνά το κόστος διοξιδίου του άνθρακα κάποια κριτήρια. Οπότε αυτό συνδυάζεται με τις εκπομπές και άλλα κριτήρια. 30 ευρώ ε, χρησιμοποίησαμε ως σημείο μία αναφορά και αυτό μπορεί να φαίνεται ψηλό ποσό για κάποιον εξωτερικό παρατηρητή. Αλλά αυτό είχαμε χρησιμοποιήσει και την περασμένη φορά, γιατί ήταν σαφέ από την οδηγία ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την τιμή τη δέσμη μέτρων ε, για το κλίμα 2020. Αυτό είχαμε κάνει και την προηγούμενη φορά. Αυτό έλεγε η οδηγία. Τώρα υπήρχαν διαφορετικέ νομικέ ερμηνείε. Έπρεπε να ακολουθήσουμε αυτή την υποχρέωση, την υποχρέωση ή να προσαρμοστούμε στα πιο πρόσφατα ε, στοιχεία. Κατά την προετοιμασία τη πρότασή μα, θεωρήσαμε ότι και δύο υποθέσει είναι βάσιμε, οπότε εκπονήθηκε αυτή η μελέτη και θεωρήσαμε ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν διαφορετικές τιμέ για τον άνθρακα, αλλά κυρίως επιμείναμε στις τιμές αυτές μαζί με άλλες, άλλα νέα στοιχεία. Και είδαμε τομεί και κλάδους με διαφορετικές τιμέ στον άνθρακα. Καταλήξαμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι τα 16,5 ευρώ μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε Όμως, ούτως ή άλλως το συμπέρασμα αυτό υπόκειται στη δυνατότητα να τροποποιηθεί ε, εφόσον τροποποιηθεί το σχετικό πολιτικό πλαίσιο. Αυτά πέρυσι. Όπως ξέρετε τον Ιανουάριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη υπέβαλε κάποιες σοβαρές προτάσεις σε σχέση με το κλίμα και την ενέργεια. Υπήρχε μια ανακοίνωση για την ενέργεια και το κλίμα με το σχετικό πρόγραμμα δράσης με στόχο το 40%. Ήταν πολύ δύσκολη η απόφαση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή και με δυσκολία συμφωνήθηκε. Θα το ξέρετε, το είπαν και κάποιοι από τους παρεμένοντε εδώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε και προτάσεις για το αποθεματικό ε, σταθερότητα τη Αγορά που μπορεί να επηρεάσει τι τιμέ του άνθρακα και να επηρεαστούν οι χαμηλέ τιμές. Αλλά συζητήθηκε πάρα πολύ και το backloading. Οπότε, από την τιμή 3,4 που είχαμε στον άνθρακα, ε, υπήρχε διαρκής το Τώρα είμαστε στο 6-7 και... και ανωδικές τάσεις. Ελπίζουμε λοιπόν η ανωδική τάση να συνεχιστεί. Αυτό ήταν το πλαίσιο όταν είδαμε την όλη πρόταση και για τον σκοπό σταθεροποίησης του σχετικού κλάδου θεωρήσαμε ότι ήταν βάσιμο να χρησιμοποιήσουν με τα 30 ευρώ ανατόνο ω τιμή αναφορά. Και ότι ήταν και νομικό ορθό στα πλαίσια τη οδηγία. Τα κράτη-μέλη, όπω είπα, συμφώνησαν σχεδόν ομοφόνο. Τώρα ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχετε την ελευθερία να αποτιμήσετε το θέμα αυτό όπω θέλετε, κάτι που κάνετε ήδη, αλλά αν αυτή η ένσταση υπερψηφιστεί θα είναι πολύ δύσκολο να σα πω τι θα γίνει. πάντω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει νέα πρόταση, διότι μπορεί να υπάρξει νέο κατάλογο όπω αναφέρθηκε, έγκριση η απουσία έγκρισης καταλόγου δεν προβλέπεται ως δυνατότητα. Απλώς θα χρειαστεί και άλλη τεχνική δουλειά και βεβαίως να προβλεφθούν πολλές συζητήσεις και πολλοί γύροι διαπραγματεύσεων. Κάτι που δεν είναι εφικτό αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να παραμείνω σε αυτά απλώ να αναφέρω το εξή. Ακούστηκε ότι λάβαμε υπόψη αυτό που συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά δεν αληθεύει. Ε, τα είδαμε πολύ προσεκτικά Είδαμε και το Λιχτενστάιν τι κάνει και άλλες ε, περιοχές για, με πολύ συγκεκριμένους καταλόγους και προσπαθήσαμε να λάβουμε τις συγκεκριμένες αποφάσεις που θεωρήσαμε ορθές. Είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω ερωτήσεις. Ο κύριος Γκρότερ. ερώτηση. Λέτε ότι δεν γνωρίζετε πόσο θα διαρκέσει. Έχουμε και τα windfall profits. Για πέστε μου, έχουμε πολλές αναλύσεις και έρευνες που γίνονται. Τι γίνεται με τα windfall profits αν δουλέψετε στη βάση των 30 ευρώ ή των 6,5 ευρώ. Μπορείτε να μας πείτε λίγο με λεπτομέρειες και να μας πείτε λίγο και το χρονικό σημείο, πιο συγκεκριμένα. Είπα ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αγοράσουν τα πιστοποιητικά του 2015 έως τον Απρίλιο 2016. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε αυτό ή μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί δεν ισχύει και πόσο θα διαρκέσει. Μέχρι τώρα χρειάστηκε πολύ καιρός μέχρι ότου καταθέσει την εξήγησή της η Κομισιόν και πρόκειται για θεμελιώδες δικαίωμα του Κοινοβουλίου που σημαίνει ότι μπορούμε να ανακόψουμε την πορεία μιας νομοθεσίας εάν δεν συμφωνούμε. Υπάρχουν πολλές αδιευκρίνιστες πτυχές. Ίσως μπορείτε ωστόσο να ρίξετε κάποιο φως σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, τα windfall profits αλλά και τι, ποιος πληρώνει τα windfall profits είναι οι καταναλωτές, αυτοί που πλέον την ενέργεια που καταναλώνουν, οι φορολογούμενοι. Μήπως μπορείτε να πείτε λίγα περισσότερα για να έχουμε κάποια συγκεκριμένα γεγονότα και, και, στοιχεία για την ψηφοφορία μας του σημερινού απογεύματο. Πρώτα ο Eichhout και μετά να επανέλθουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει. Και εγώ έχω μερικές ερωτήσεις προς την Κομισιόν κύριε Πρόεδρε διότι δεν ήταν ας πούμε σαφής όλες οι απαντήσεις που έδωσε. Είπατε ότι έχει αλλάξει το πολιτικό ας πούμε πρόγραμμα. Μέσα στην μελέτη αντικτύπου λαμβάνετε υπόψη το backloading στην ανάπτυξη των ε, ε, τιμών σας. Στο VK33 βλέπετε να περιλαμβάνονται οι τιμές, περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς. Δεύτερο, οι προτάσεις για τις οποίες μιλείτε, το πακέτο 2030 για παράδειγμα, αρχίζουν όλες το 2021. Ενώ τώρα εμείς μιλούμε για μια λίστα μέχρι το 2020. Να πούμε λοιπόν σωστά τις χρονολογίες. Υπάρχουν νέες προτάσεις, αλλά αυτές αρχίζουν να εφαρμόζονται μετά το 2020. Και εμείς μιλάμε εδώ για τη λίστα διαρροής του άνθρακα μέχρι το 2020. Για να τα ξεκαθαρίσουμε. Δεύτερο, είπατε ότι τεχνικά χρειαζόμαστε χρόνο για να φτιάξουμε νέα λίστα carbon leakage. Και χαίρομαι που είπατε ότι θα καταρτήσετε νέα λίστα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Όμως ήσασταν λίγο ασαφείς σχετικά με το πόσο θα χρειαστεί για να γίνει αυτό. Διότι περιλαμβάνουμε ήδη τις πολιτικές συζητήσεις. Αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει τώρα αυτό, διότι δεν είναι και δική σας υπόθεση αυτή για την ώρα. Τεχνικά μπορείτε να κάνετε λίστα και αύριο. Διότι στην μελέτη αντικτύπου έχετε ήδη υπολογίσει τις εξοικονομήσεις ή το πρόσθετο εισόδημα αν πάρετε 6,5 ευρώ αντί 30. Είναι λοιπόν πολύ ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα μέσα στη μελέτη αντικτύπου. Άρα πρέπει η λίστα να είναι σχεδόν έτοιμη. Τεχνικά λοιπόν μπορείτε να την φτιάξετε ταχύτατα. Και θα ήθελα να μου πείτε, πολιτικά είναι άλλη υπόθεση. Αυτό είναι βέβαια υπόθεση των πολιτικών ανδρών και γυναικών. Αλλά τεχνικά πόσο χρόνο σας χρειάζεται Τελευταία παρατήρηση για τα επιχειρηματικά λόμπι για τους συναδέλφους εκείνους οι οποίοι ανησυχούν για τα 30 ευρώ. Κάθε φορά που θα συζητούμε αναθεώρηση του συστήματος ETS και που θα πείτε μην το αγγίζετε το σύστημα, θυμηθείτε ότι τα λόμπι λένε ότι κάνουμε τον υπολογισμό ήδη με τα 30 ευρώ. Όταν μιλούσαμε όμως για το backloading μας είχαν πει είναι πρόβλημα για μας να πάμε από τα 5 στα 6 ευρώ. Α, και τις επενδύσεις όμως μιλούμε για 30 ευρώ. Α, τελικά business τι χρησιμοποιείτε, τα 30 ευρώ ή τα 5 ευρώ. Σταματήστε λοιπόν τις ανοησίες. Και η πολιτική να είμαστε ευφυείς και τα λόμπι να είναι συνεπέστερα, διότι χρησιμοποιούν οποιοδήποτε επιχείρημα, με οποιοδήποτε τρόπο, όταν θέλουν να μας πείσουν. Λοιπόν, να δούμε ακριβώς πού στοχεύουν τα επιχείρηματά τους. Τώρα η Επιτροπή, λέει ο Πρόεδρος, δηλαδή η Κομισιόν. Κοιτάξτε, ποιος κερδίζει και ποιος χάνει αν γίνει συντομότερος ο κατάλογος. Έχουμε κάνει κάποιες υποθέσεις μικρότερη λίστα, μικρότερες free allocations σε ορισμένους τομείς, άρα περισσότερες allowances που θα μπουν σε πληστηριασμούς στο μέλλον. Και το εισόδημα αυτό θα καταλήξει στις χώρες μέλη. Σε αυτό συμφωνείτε νομίζω, γιατί συμφωνείτε με τη μελέτη αντικτύπου. Είπαμε ότι αυτός ο διορθωτικός παράγοντας, ο διορθωτικός συντελεστής θα επανυπολογιστεί και ίσως θα πάει τελικά σε αυτούς που θα παραμείνουν στη λίστα. Αλλά αυτό δεν είναι σίγουρο. αν υπάρχει λιγότερη δωρεάν allocation σε ορισμένους τομείς βιομηχανίας θα περάσει το κόστος και ίσως τα προϊόντα να, είναι, να μην είναι τόσο ακριβά. Ή θα γίνουν τα προϊόντα φθηνότερα και τότε θα χάσουν οι μέτοχοι. Όλα αυτά τέλος πάντων είναι διαφορετικά ανάλογα με την επιλογή που θα κάνει κανείς και είναι, δεν έχει υπολογιστεί ακόμα από όλες τις επιχειρήσεις πώς. Βεβαίω και μπορείτε να απορρίψετε την ε, λίστα. Δικαίωμά σας είναι. Για το timing. Στην πράξη όντως έχουμε όλα τα δεδομένα και μπορούμε να συντάξουμε την νέα λίστα πολύ σύντομα. Αλλά οφείλω να υπογραμμίσω ότι στην οδηγία προβλέπεται η συμπερίληψη και κριτηρίων ποιότητος που είναι πιο χαλαρά. Έχουμε διάφορους τομείς τώρα που δεν ήταν στη λίστα αρχικά βασισμένη στα νούμερα, αλλά βασισμένη σε αυτά τα κριτήρια ποιότητα. Και αυτό που μπορούμε να προβλέψουμε είναι ότι αν είναι συντομότερο ο κατάλογο, θα ληφθούν περισσότερο υπόψη τα κριτήρια ποιότητα. Και αυτά χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Αυτό είναι ένα στοιχείο αβεβαιότητας που υπησέρχεται. Eichhout είπε ότι το backloading έχει περιληφθεί σε ορισμένες από τις προβλέψεις τιμών. Αυτό είναι σωστό. Και συμφωνώ μεν ότι το MSR και ότι είναι πιο σαφή για τα μετά το 2020 τίθεται σε κίνδυνο η αξιοπιστία του ETS. Ήταν αλλιώ τα πράγματα πριν που ήταν πολύ χαμηλή αξιοπιστία του ETS και είναι αλλιώ τα πράγματα σήμερα. Ελπίζω να σα απάντησα. Ευχαριστούμε. Νομίζω κάναμε μία πλήρη συζήτηση από το σημείο αυτό. Ίσως οι ομάδες να μπορούν μετά να δουν με μεγαλύτερη προσοχή πώς βλέπουν τις διάφορες τοποθετήσει. Να σας πω ότι θα αποφασίσουμε και θα ψηφίσουμε όταν συνεχιστεί η συνεδρία στο απόγευμα και τώρα θα έχουμε την κοινή συζήτηση στα σημεία 7 και 8 ένσταση βέσου του 106 κανονισμό της Επιτροπής για την κατάσταση του παράρτηματος 3 της οδηγίας 2008-98 ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα και την κατάρριξη ορισμένων οδηγιών. Και επίσης μαζί με το σημείο 8 και πάλι ένσταση βάση του άρθρου 106 απόφαση της Επιτροπής που προβοποιεί την απόφαση 2532 ΕΚ σχετικά με τον κατάλογο των αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2898. Και για τις δύο περιπτώσεις θα δώσω το λόγο στη συνάδελφο Κέστιγκερ η οποία ε, έχει προβάλλει την ένσταση και μετά θα έχουμε μια ολόκληρη συζήτηση για να ακούσουμε τι απόψει όλων των πολιτικών ομάδων. Παρακαλώ, Ελίζαμπετ. Ähm, äh, Ευχαριστώ. Σύντομα για τις ενστάσεις ε, θα τις συζητήσω και δυο μαζί. Πρώτη ενστασία. για την προσαρμογή στο classification leveling και τα λοιπά των μήλων. Για την πρώτη ένσταση υπάρχει πρόβλημα με την τροποποίηση του παραρτήματος 3, διότι τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά εδώ περιγράφονται πολύ ασαφώς σε σχέση με κανονισμούς που ήδη ισχύουν στις χώρες μέλη. Επίσης δεν έχουν οριστεί οριακές τιμές και διαδικασίες εξετάσεως, κάτι το οποίο δίνει, κάνει δύσκολο να εφαρμοστούν οι διατάξεις του κανονισμού και το κριτήριο του κινδύνου, το οικοτοξικό, έχει μείνει απ' έξω από το κείμενο του κανονισμού. Και παραμένει στην ευχέρεια των ε, χωρών μελών. Τέταρτο, η αλλαγή του κριτηρίου επικινδυνότητας HP4. Εδώ μπορούν να υπάρξουν προβλήματα σε σχέση με την χρήση υπολείπων καύσεως από ξύλο ή τύρφη κλπ που μπορούν να έχουν οξύδια ή υδροξίδια του ασβέστου και που χρησιμοποιούνται μετά στην, ε, ως λιπάσματα. Δεύτερη ένσταση για τροποποίηση του χαρακτηρισμού των μήλων. Εδώ περιλαμβάνονται τρεις νέοι χαρακτηρισμοί. Πρώτον, ο μεταλλικός υδράργυρος σταθεροποιητικός υδράργυρος και τρίτο ερυθρά υλής. Αυτά το μεταλλικό σιδάργυρος και ο εν μέρη σταθεροποιημένος σιδάργυρος δεν ήταν απαραίτητα διότι έχουν ληφθεί υπόψη τα κατάλοιπα αυτά υδαργύρου στα ε, διάφορα, στη διάφορα νομοθετήματα που υπάρχουν ήδη. Αυτό σημαίνει δηλαδή ε, ε, δεν είναι δυνατόν να διαβάζει τόσο γρήγορα η κυρία Κέστιν και, να επιμένει να τη μεταφράσουμε κιόλα. Είναι πάρα πολύ τεχνικό το δέχεται κύρια. Λοιπόν δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι κωδικοί αυτοί. Το πρόβλημα είναι λοιπόν ότι υπάρχει επικάλυψη και υπάρχουν και διαφορετικές διατάξεις στις χώρες μέλη. Αυτά και πολύ σύντομα, διότι βέβαια το θέμα είναι πάρα πολύ περίπλοκο και τεχνικό και θα ήθελα να ακούσω τώρα τις απαντήσεις της Επιτροπής. Grazie. Σας ευχαριστούμε. Η ε, συνάδελφος Μάισνερ απλώς έχει ζητήσει το λόγο. Να τη δώσω αμέσως το λόγο. Ε, κυρία Μάισνερ, ευχαριστώ. Τα άκουσα αυτά. Η ομάδα των φιλελευθέρων δεν δέχεται την ένστασή σας διότι θεωρούμε ότι οι νέες νομοθετικές προτάσεις είναι μάλιστα φιλικότερες για τους καταναλωτές. Χρειάζεται, είπε και η κυρία κυρία Κωστινγκέ, περισσότερο χρόνο. Τον χρόνο αυτό δεν τον έχουμε όμω. Η Αυστρία επιθυμεί να ζητήσει κάτι το νέο, ναι, οι άλλε όμω χώρε όχι. Το ζήτημα είναι, είναι σκόπιμο αυτό. Αυτά είναι τεχνικέ λεπτομέρειε, πολύ τεχνικέ και νομίζω πρέπει να τα αφήσουμε στα χέρια των εμπειρογνωμόνων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι συνάδελφοί μου δεν βλέπουν κανένα λόγο στην πολιτική μου ομάδα δηλαδή να εγείρουμε ένσταση. Οι προσαρμογέ θα πρέπει να γίνουν στι εθνικέ νομοθεσίε. Αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται και επανέρχεται. Τα εξετάσαμε αυτά εκ του σύνεγγυ, αλλά νομίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να συνεχίσει με τη διαδικασία αυτή και εμείς πάντως δεν πρόκειται να δεχθούμε την ένσταση. Ευχαριστώ. Εάν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, να δώσω το λόγο ευθύ αμέσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας απαντήσουν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι ο Χούλιο Καρθιά που είμαι επικεφαλής του τμήματος ε, που ασχολείται με το θέμα των ε, αποβλήτων στην σχετική γενική διεύθυνση και επιτρέψτε μου να κάνω κάποιες προκατρακτικές παρατηρήσεις. Να πω ότι τα δύο σχέδια κανονισμού για τον κατάλογο των αποβλήτων και την κατάργηση των οδηγιών δεν εμφανίστηκαν από το πουθενά. Είναι κατάληξη μιας εργασίας που κράτησε μια πενταετία με πολλαπλές συζητήσεις επιδογνωμόνων, επανειλημμένες συνεδριάσεις επιτροπών, τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών και πάρα πολλές τεχνικές πληροφορίες. Η τεχνική πολυπλοκότητα του θέματος είναι τεραστία. Αλλά Χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι τα περισσότερα ενδιαφερόμενα μέρη στηρίζουν τα σχέδια των κανονισμών και ότι στην Επιτροπή για τα Απόβλητα υπήρξε μια σαφή τοποθέτηση της πλειοψηφία των κρατών μελών υπέρ της ε, νομοθεσίας αυτής. Είχαμε 24 ε, θετικές ψήφους και για τους δύο κανονισμούς και μόνο τρία κράτη-μέλη, η Αυστρία, η Ελλάδα και η Πολωνία κατεψήφισαν για διαφορετικούς βεβαίως λόγους. Και τώρα θα διατρέξω τα επιχειρήματα που προέβαλε η κυρία Κέστιγκερ. Είναι πραγματικά τεχνικός πολύπλοκο το θέμα και είναι σημαντικό η Επιτροπή σας να έχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στη διάθεσή της. Η παρέμβασή μου λοιπόν θα είναι και μακροσκελέστατη και λεπτομερέστατη και περισσότερο το βορτέρων. Συγγνώμη γι' αυτό. Πρόεδρε, στην πρόταση ψηφίσματος υποβλήθησαν τρία διαδικαστικά επιχειρήματα. Πρώτα απ' όλα ότι υπερεύει την ετολή της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του παρατήματος 3 της οδηγίας για τα απόβλητα και παρά τα τεχνικά και επιστημονικά στοιχεία. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε αυτό συμφώνησε η Επιτροπή για τα απόβλητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε να κάνει κάτι ακόμη πιο αυτόματο από μια τεχνική προσαρμογή. Ευθυγραμμίζουμε τις ιδιότητες προβλέπονται στην νομοθεσία για τα απόβλητα με αυτές τις χημικής της για τα χημικά. Για τα, χημικά. Η, τα χαρακτηριστικά αυτά αναφέρονται πλέον στον κανονισμό του 2008 για την ταξινόμηση και την επενσήμαση και τη συσκευασία των χημικών ουσιών και ο κανονισμός αυτός ουσιαστικά αντικατοπτρίζει την τεχνική και επιστημονική σχετικά πρόοδο, ευθυγραμμίζοντας την χημική νομοθεσία με το σύστημα ε, ταξινόμησης των χημικών ουσιών του ΟΗΕ. Σε μια δεύτερη φάση να πω ότι η Επιτροπή αποβλήτων ότι είμαστε μία και μόνη γνωμοδότηση για τα δύο σχέδια κανονισμών. Όμως Φοβούμε ότι το επιχείρημα αυτό δεν ε, βαρύνει διότι όντως η Επιτροπή ετοίμασε δύο γνωμοδοτήσεις, υπήρχαν δύο κατάλογοι ψηφοφοριών και στο μητρό της Επιτροπολογίας δύο διαφορετικές καταχωρήσεις. Ε, ψηφίστηκαν λοιπόν ξεχωριστά οι δύο προτάσεις, αλλά επειδή είναι πραγματικά πολύ στενά συνδεδεμένες να αναφέρονται από κοινού. Δεν υπήρξαν μάλιστα καθόλου αντιρρήσεις, ούτε καν από αυτούς που κατεψήφισαν για τον κατάλογο. Οπότε νομίζω ότι αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε και μια κοινή συζήτηση σήμερα, έτσι. Επί της ουσίας, Ακούστηκε το επιχείρημα ότι οι ορισμοί στο σχέδιο των κανονισμών είναι ασαφεί, ανοιχτέ ερμηνεία και θα δημιουργήσουν νομική βεβαιότητα. Ωστόσο, οι επικίνδυνε ουσίε τώρα ορίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια ε, στα σχέδια κανονισμών από ό,τι στο παρελθόν. Μάλιστα, η δήλωση περί κινδύνων και τα σχετικά παραθέματα αυξάνουν την νομική βεβαιότητα. Έπειτα ακούστηκε το επιχείρημα ότι ο ορισμός επικίνδυνη ουσία σημαίνει ότι πολλά απόβλητα, ιδίως στο κατασκευαστικό τομέα ή τα παράγωγα της αποτέφρωσης, θα πρέπει να είναι ταξινομημένη η επικίνδυνη ουσία. Δεν είναι αυτή όμως περισχύουσα άποψη μεταξύ των ειδικών και μάλιστα πλειοψηφία των κρατών μελών της Επιτροπής Αποκλήτων δεν δέχτηκε αυτή την ένσταση. Σε κάθε περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποσαφηνίσει το όλο ζήτημα και μέσω των εγγράφων που σκοπεύουμε να δημοσιεύσουμε θα διευκρινίσουμε ποια είναι τα απόβλητα που είναι επικίνδυνα ή μπορεί να δημιουργούν άλλου είδους ε, ρήπανση ακριβώς μέσα από τη διαδικασία της απανθράκωσης. Το σχέδιο κανονισμού δεν προβλέπει, λέγεται, ορισμό για την επικίνδυνη ουσία 14, την εκοτοξίνη. Όμως, αυτό καλύπτεται και δεν υπάρχει νομικό κενό εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, φροντίζει να εκπονηθεί μελέτη για το θέμα αυτό, την επικίνδυνη ουσία 14. Άλλωστε, στο σχετικό σχέδιο ψηφίσματος λέγεται ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν τη σχετική τους νομοθεσία δις και αυτή τη φορά και τώρα δηλαδή και αφού ολοκληρωθεί η αποτίμηση για την επικίνδυνη ουσία 14. Όμως είναι δύσκολο να γίνουν κατανοητά τα επιχειρήματά σας τώρα διότι η πρόθεσή μας ακριβώς ήταν να προσαρμόσουμε τον κανονισμό. Τον κανονισμό που εφαρμόζεται αυτομάτως και δεν απαιτεί κανενός είδους μεταφορά. Το σχέδιο ψηφίσματος υπάρχει και μια αντίρρηση για το ότι δεν δημοσιεύτηκε η μελέτη αντικτύπου. Είναι και αυτό επί διαδικαστικού αντίρρηση, αλλά να τονίσω και να επισημάνω ότι τέτοια μελέτη αντικτύπου δεν ε, απαιτείται για μέτρα επιτροπολογίας και η νομοθεσία για το διοξίδιο του άνθρακα βάσει της οποίας ελήφθη η δική μας απόφαση βασίστηκε σε πρόσθετα επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία βάση των απόψεων που κατέθεσαν και τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως είπα σε μια δουλειά πενταετίας. Στο σχέδιο κανονισμού τώρα για την ε, τροποποίηση του καταλόγου κατανόησα τη βασική αντίρρηση στο σχέδιο ψηφιακού, στην ένσταση δηλαδή, που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να έχει μια ριζοσπαστικότερη προσέγγιση στον κατάλογο των αποβλήτων. Η αντίρρηση αφορά τη μελέτη που εκπονήθηκε το 2008 για, μια πλήρως, για έναν τελείως νέο κατάλογο αποβλήτων. Όταν καταλήξαμε σε αυτή τη μορφή ήταν σαφές ότι οι εθνικές αρχές και οι ενδιαφερόμενοι δεν ήθελαν ριζοσπαστικές αλλαγές απλώς και μόνο διότι το κόστος της προσαρμογής σε έναν τελείως νέο κατάλογο, ακρεφνός καινούριο, θα ήταν πολύ σοβαρό. Ε, κατά τα άλλα, θεωρώ ότι τα επιχειρήματα που ε, προβάλλονται στο κοινό της ένσταση δείχνουν κάποια έλλειψη κατανόησης για το πώς λειτουργεί η νομοθεσία για τα απόβλητα στην πράξη. Υπάρχουν κάποια απόβλητα για τα οποία υπάρχουν απόλυτα αριθμητικά στοιχεία, αλλά ο εντοπισμό των αποβλήτων που θα θεωρηθούν επικίνδυνα ή μη είναι κάτι πολύ σοβαρό. Έπειτα έχουμε τις λεγόμενες mirror entries, δηλαδή τις καταχωρήσεις ε, κατά προσέγγιση, όπου αναπερίπτωση υπολογίζουμε τα απόβλητα και ε, από τον όγκο καθορίζεται επικινδυνότητα και επίσης υπάρχει και μια πολύ μεγάλη ευελιξία στην ε, δομή του συστήματος. Η ευελιξία αυτή επιτρέπει στα κράτη-μέλη μερικά πράγματα να μην τα θεωρούν επικίνδυνα απόβλητα Αυτό σημαίνει ότι εισάγονται νέα στοιχεία στο σύστημα και διατηρούνται σύμφωνα με όλες ε, τις χώρες μέλη. Μόνο η Αυστρία θέλει το βασικό σχεδιασμό. Δεν ξέρω τι σύστημα θέλει να καθορίσει η Αυστρία. Αυτό όμως που είναι σαφές για μένα είναι ότι οι διαρθρωτικές αλλαγές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν οικονομικές και περιβαλλοντικές δυσκολίες. Τέλος, άλλο επιχείρημα είναι ότι οι νέες ιδιώτες επικινδύνων δεν λαμβάνονται υπόψη στην τροποποίηση του καταλόγου αποβλήτων. Και δίνεται το παράδειγμα σύμφωνα την πρόταση ψηφίσματος οι μπαταρίες που θα έπρεπε να ταξινομούνται ως επικίνδυνες ουσίες. Όμως η ανάλυση που έγινε πριν από την τροπολογία δεν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αναθεώρηση βάσει αυτού θα είχε κάποιες επιπτώσεις στον κατάλογο των επικινδύνων. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση των ε, μπαταριών πρέπει να σας πω ότι σήμερα ήδη έχουν μία ή δύο από τις ιδιότητες των επικινδύνων, προβλέπεται δηλαδή αυτό. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη συμφωνήσει να προχωρήσει σε αναθεώρηση του περιεχομένου, ξεκινώντας μάλιστα από τις μπαταρίες και συζητώντας επ' αυτού με τα κράτη-μέλη. Αν κατακλείδη, Πρόεδρε, θέλω να ζητήσω από την Επιτροπή σας να μην στηρίξει τις δύο ενστάσεις Πρώτον, διότι πιστεύουμε ότι τα δύο σχέδια κανονισμού είναι σαφή και αποτελούν σαφή βελτίωση σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση. Δεύτερον, εάν περνούσαν οι ενστάσεις, τότε θα αντιμετωπίζαμε μία κατάσταση ασυνέπειας στην ομοθεσία μας γιατί δεν θα υπήρχε συνέπεια να, με τον κανονισμό CLP, ο οποίος εφαρμόζεται πλήρως από του χρόνου βάσει της οδηγίας ε, για την εισαγωγή αποβλήτων. Και τρίτον, γιατί δεν θα μπορούσαμε έτσι να συμμορφωθούμε με τις διεθνείς μας υποχρεώσεις βάσει της ε, σύμβασης για τον υδράργυρο. Εξού και η πρότασή μας, η οποία έχει σαν στόχο να διασφαλίσει ότι τα πόβλητα υδραργύρου θεωρούνται επικίνδυνα. Όπως και να έχει το πράγμα πάντως, μπορώ να σας διαβεβαιώσω για το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να κάνει περισσότερα πράγματα και να εκδώσει οδηγίες προκειμένου να διασφαλίσει εναρμονισμένη εφαρμογή του καταλόγου αποβλήτων με επικίνδυνες ιδιότητες. Αναμφίβολα θα συνεχίσουμε και το έργο μας όσον αφορά την τοξικότητα και την επικινδυνότητα των ε, προϊόντων μεταξύ άλλων και των μπαταριών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίασή της αυτή και για τις επεξηγήσεις που μας έδωσε σε βάθος. Με το σημείο αυτό δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι έχουμε τίποτα άλλο στην ημερήσια διάταξη και σήμερα το πρωί. Οπότε στις 3 το απόγευμα θα ξαναβρεθούμε για να συνεχίσουμε τις εργασίες μας.